Καθίστε παρακαλώ συναδελφοί, παρόλο που δεν είναι ασφιχτικά γεμάτη η αίθουσα, ε, ε, έχουμε περιορισμένο χρόνο, καλό θα ήταν να αρχίζαμε και να περάσουμε αμέσως στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης με θέμα επισκόπηση του πιλωτικού προγράμματος 2015-2016 δοκιμαστικό σχέδιο ήταν αυτό και μετά προπαρασκευαστική δράση για την περίοδο 2017-2019. Έχει έρθει η ώρα του απολογισμού να δούμε ε, τι έχει γίνει και ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον. Και με χαρά και τιμή θέλω να καλωσορίσω δύο μέλη Mrs. του πάνελ είναι η κυρία Σίλβια Κάιντς Χούμπερ, ε, τμήματάρχη στη Γενική Διεύθυνση Grow, ε, ε, το τμήμα 15 για την άμυνα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τον κύριο Dirk Tilburger, ο οποίος είναι αναπληρωτής διευθυντής για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Αφιερώνουμε εμείς αρκετό χρόνο σήμερα στη συζήτηση και για τα δύο θέματα. Οπότε δεν χρειάζεται εγώ να μακρηγορήσω. Και θέλω να δώσω μέσα στο λόγο στην κυρία Κάιντς Χούμπερ, πρώτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στον κύριο Μπέρκερ. Κύριε μου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν περάσουμε στην παρουσίαση των συγκεκριμένων έργων που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί ή που προετοιμάζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια εισαγωγικά και το ε, ιστορικό και για το πιλωτικό πρόγραμμα και για την προπαρασκευαστική δράση. Ε, ήταν και τα δύο για την έρευνα στην αμυντική βιομηχανία με στόχο να βολιδοσκοπήσουμε τις δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για ε, κοινά προγράμματα έρευνας. Ε, το πιλωτικό πρόγραμμα αυτό και η προπαρασκευαστική δράση και τα δύο ε, ανατέθηκαν ως προς το εφαρμοστικό σκέλος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος από ένα ε, προηγούμενο πιλωτικό πρόγραμμα που ήταν το αρχικό και σε μικρή κλίμακα. Και πώς έγινε ο επιμερισμός εργασίας. Ε, εκείνη τη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να καταθέσει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα εργασίας. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση ποιών έργων αλλά ε, με πρόταση του προγράμματος εργασίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Και στη συνέχεια στην προπαρασκευαστική δράση ε, για την αμυντική έρευνα ολοκληρώθηκε αυτή η φάση από το 17 μέχρι το 19. 90 εκατομμύρια είναι ο συνολικός ε, προϋπολογισμός με στόχο να βολιδοσκοπήσουμε ακριβώς αυτό, πώς μπορεί να χρηματοδοτήσει η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση κοινά προγράμματα συνεργασίας για την άμυνα. Full scale και στο μέλλον να γίνει ένα πλήρες πρόγραμμα που προτείνεται, από το, ε, που είναι το Ευρωπαϊκό Ταμιντικό Ταμείο και να ε, δοκιμάσουμε και τους μηχανισμούς που μπορούν να οδηγήσουν εκεί. Συμφωνήσαμε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να του αναθέσουμε αυτό το έργο Ακριβώς πάλι σε συνεργασία επιμερίζεται το έργο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει το πρόγραμμα εργασίας σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Συστήνεται ομάδα εμπειρογνωμόνων που μας υποστηρίζει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας εκεί είναι παρατηρητής σε αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Μας δίνει ενημέρωση εκ των προτέρων και εκ των υστέρων για διάφορα ερευνητικά προγράμματα και θέματα σε σχέση με το σχέδιο ανάπτυξη δυναμικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια εγκρίνει αυτό το πρόγραμμα εργασίας. που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ε, τα κείμενα προκήρυξη των διαγωνισμών. Και αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί αυτό, παραδίδεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας που προκυρεί στο διαγωνισμό, κάνει την αξιολόγηση, ε, προετοιμάζει τις συμφωνίες χρηματοδότησης και όταν αυτές υπογραφούν ε, παρακολουθεί και την εκτέλεση του έργου. Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η διαδικασία και ο τρόπος ε, με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για την προπαρασκευαστική δράση. Το πρόγραμμα εργασίας, σας είπα, είναι σε αιτήσια βάση και καταρτίζεται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Στην αρχή χονδρικά και πάλι μαζί με τα κράτη-μέλη και μετά από προτάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας αλλά και άλλων ενδιαφερομένων εντοπίσαμε τέσσερα μεγάλα είδη ερευνητικής δραστηριότητας. Θέλαμε να έχουμε προγράμματα επίδειξης, ε, ασχοληθούμε με κρίσιμες ε, αμυντικές τεχνολογίες, ε, έρευνα για το μέλλον και αναδυόμενες τεχνολογίες που ανατρεπτικές. Παράλληλα, έχουμε εντοπίσει και τέσσερις μεγάλους τομείς δραστηριοτήτων Σύφορα εσα προταση ε, προστασία των δυνάμεων και πλατφόρμες μη επανδρομένες. Συνδυάσαμε λοιπόν όλους αυτούς τους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τα τρία ετήσια προγράμματα εργασίας που ε, προετοιμάζουμε στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής αυτής δράσης. Βρισκόμαστε τώρα, διανύουμε το τρίτο έτος μας. Το πρώτο πρόγραμμα εργασίας για το 2017 και το δεύτερο για το 2018 προφανώς ήδη έχουν εγκριθεί αλλά και εφαρμοστεί, εκτελεστεί, έχουν γίνει διαγωνισμοί και τα έργα από τους διαγωνισμούς του Εφτά έχουν ήδη υπογραφεί και τρέχουν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια την περιγραφή και από, την προκήρυξη του διαγωνισμού την περσινή του Μαρτίου. Τελειώνει η αξιολόγηση αυτό τον καιρό, είναι στο τελικό στάδιο, στα τελευταία βήματα με τις συμφωνίες χρηματοδότησης για τα διάφορα έργα που επίκειται η υπογραφή τους, ελπίζω ακόμα μέσα στο Μάρτιο. Και έχουμε και ένα τρίτο πρόγραμμα εργασίας τώρα, για το 19 που είναι το τελευταίο στη συγκεκριμένη προπαρασκευαστική δράση, έχει ολοκληρωθεί και είναι στη διαδικασία έγκρισης. Και επίσης έχουμε εγκρίνει και θέλουμε, μάλλον ιδανικά να υιοθετηθεί με το νέο πρόγραμμα εργασίας για το EDIDP. από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και το σκέλος της ανάπτυξης. Να μπω λίγο και σε κάποιες στατιστικές. Πρόγραμμα εργασίας του 2017 εστίασε σε τρεις μεγάλους διαγωνισμούς για τα μη επαδρομένα συστήματα. Είναι ένα πρόγραμμα επίδειξης υψηλής ε, ορατότητας και προβολής που θα σας παρουσιάσει ο επόμενος ομιλητής. Ε, προστασία των δυνάμεων και των ε, στρατιωτών και το τρίτο ήταν μια προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ε, τη μελλοντική τεχνολογία για να δούμε ποιες είναι οι κρίσιμες τεχνολογίες για την άμυνα στο μέλλον. Στατιστικές γενικά από τους τρεις διαγωνισμούς ήταν με ένα προπολογισμό 43 εκατομμύρια και κάτι, 21 προτάσεις καταθέθηκαν. ...147 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε. 447 ζήτησαν, ε, ζητούσαν τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και άλλοι ενδιαφερόμενοι τμήματα του ομίλου. 187 συνολικά ε, ήταν οι διάφοροι συμμετέχοντες. Πέντε έργα χρηματοδοτήσαμε ε, από το διαγωνισμό αυτό. Και διαπιστώσαμε επίσης ότι η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν καλή, ιδιαίτερα για τα συστήματα προστασίας των στρατιωτών. Και αυτό που προσπαθούμε είναι να ισορροπήσει κάπως το πρόγραμμα εργασίας. Δηλαδή να έχουμε και διαγωνισμούς που να προσελκύουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτός από τις γνωστές ε, των μεγάλων πέντε κρατών μελών που έχουν και τη μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη, Ιταλία, δηλαδή Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Έχουμε και μικρομεσαίες από τις κάτω χώρες, την Πολωνία, την Εστονία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο κλπ. Πάρα πολύ γρήγορα για το δεύτερο διαγωνισμό για τον ηλεκτρονικό ε, σχέδιο και λέιζερ υψηλής ε, ε, ισχύως. και επίσης για τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Είναι διαφορετικές εδώ οι στατιστικές. Επτά ήταν οι αιτήσεις που κατατέθηκαν. Για ποιο λόγο. Ε, ήταν πάρα πολύ ειδικά τα θέματα αυτή τη φορά. Γι' αυτό ε, ασχολούμαστε με τις κρίσιμες τεχνολογίες για την άμυνα, ε, όπου είναι και λιγότεροι συμμετέχοντες και εκείνοι που θα υποβάλουν αίτηση. Ήταν κάποιοι όμιλοι ε, που πληρούσαν τα κριτήρια Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό και ο προπολογισμό γενικά ήταν ε, χαμηλότερο, 19,3 εκατομμύρια για το 2018. Επίση, ε, σε αυτά τα έργα ή στις προτάσεις μάλλον, αυτά που ζητούσαν ήταν, ε, ήταν 85 οι συμμετέχοντες. Τελικά χρηματοδοτήσαμε τρία έργα και παρόλη την ιδιαίτερη υφή και χαρακτήρα του προγράμματος ήταν μόλις το 24% η συμμετοχή. Αυτή η προπαρασκευαστική δράση λοιπόν απέδωσε, ε, ε, προσέλκυσε το ενδιαφέρον και της βιομηχανίας και των ερευνητικών κέντρων και πραγματικά ε, θα πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως και δρομολογήθηκαν συνεργατικά προγράμματα σε αυτή την προπαρασκευαστική δράση. Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή για την αμυντική έρευνα. Τελευταίο, πώς επιλέγονται τα έργα. Γιατί αυτό ε, γέννησε πολλά ερωτηματικά. Πώς επιλέξαμε τα έργα. Εμείς βασιστήκαμε σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έκαναν την αξιολόγηση και στη συνέχεια προκηρύχθηκε διαγωνισμός, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να επιλέξουμε ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων από διάφορα κράτη-μέλη με διαφορετική πραγματογνωμοσύνη και γνώσεις ο καθένας για να μπορούν αποτελεσματικά να αξιολογήσουν διάφορες προτάσεις και διάφορες ε, προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Χρειαζόταν και κάποια άδεια ε, για να έχουν πρόσβαση σε ε, διαβαθμισμένα έγγραφα και βεβαίως δεν έπρεπε οι εμπειρογνώμονες να έχουν σύγκρουση συμφερόντων ή καμία σχέση με τα προγράμματα ή τις αιτήσει που εκλήθησαν να αξιολογήσουν. Τα κριτήρια ήταν τα ίδια που χρησιμοποιούμε με την έρευνα για πολιτικούς σκοπούς. Ε, αριστεία, αντίκτυπος, ε, εφαρμογή του προγράμματος, ε, το οποίο έργο κάθε φορά μπορεί να σπάσει και σε πιο μικρά κομμάτια ανάλογα με τα ειδικά κριτήρια της απαιτήσει του. Και κάτι άλλο που θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε, ε, που το κάνουμε έτσι και αλλιώς και το εφαρμόζουμε και στην προπαρασκευαστική δράση, είναι ένας δεοντολογικός έλεγχος. Δηλαδή, κάποια έργα που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, στη συνέχεια περνούν από ένα δεοντολογικό έλεγχο για την εφαρμογή και εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων. Γίνονται συστάσεις στη συνέχεια, ε, τα οποία ε, οι συστάσεις αυτές αναφέρονται στις συμφωνίες χρηματοδότησης με τους ομίλους. Και πριν υπογραφούν οι συμβάσεις, γίνεται και ένας έλεγχος ασφαλείας. Δηλαδή, βάσει των συστάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, των χωρών από τον οποίο προέρχονται τα μέλη του ομίλου, καλούνται αυτές οι χώρες να μας βοηθήσουν να κάνουν συστάσεις για τον έλεγχο ασφαλείας και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία του προγράμματος, κάποια αποτελέσματα που περιμένουμε θα πρέπει να ε, είναι διαβαθμισμένα. Και ακολουθείται η συνήθις διαδικασία τα, από τις προτάσεις και τις συστάσεις των εμπειρογνωμών. Θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Thank you for your time. Σας ευχαριστώ. Give the floor to Mr. Ο κ. Dirk Tilberger, αναπληρωτής διευθυντής στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην υποεπιτροπή σας για τα πιλωτικά προγράμματα και την προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον αμυντικό χώρο. Θα σας εξηγήσω ποια είναι τα πιλωτικά προγράμματα και ποια είναι η προπαρασκευαστική δράση που εστιάζουν σε τρία project. Το ένα είναι πιλωτικό, τρία είναι όλα όλα. Το μεγαλύτερο project ε, της προπαρασκευαστικής δράσης είναι τεχνολογικής υφής και το άλλο είναι για την προστασία των ε, στρατιωτών, συστήματα προστασίας στρατιωτών. Επέλεξα ένα project για να σας μιλήσω λίγο περισσότερο γι' αυτό. Θα μπω λίγο σε λεπτομέρειες σε αυτά τρία project, τι κάνουμε ακριβώς με αυτά, τι προωθούμε. Το πιλωτικό καταρχάς ε, σχέδιο Βλέπετε το χρονοδιάγραμμά του. Ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση το 2015-2016, η προπαρασκευτική δράση το 2017 μέχρι το 2019 και όλα αυτά ε, φυσικά ετοιμάζουν το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, υπό το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Ε, μιλάμε τώρα για μια συμφωνία εκχώρησης που υπογράφηκε το, 16 Νοεμβρίου του 2015 και εμείς στον αμυντικό οργανισμό ε, είμαστε υπεύθυνοι για το πιλωτικό πρόγραμμα και τις ε, δράσεις του. Ε, η προκήρυξη διαγωνισμού έγινε, έγινε η αξιολόγηση και η συμφωνία για τη χρηματοδότηση, όλα αυτά με συντονισμό του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού. 1,4 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προπολογισμό, μικρό προπολογισμό, θαυμάσια όμω αρχή για το, τη χρηματοδότηση τη έρευνα στον τομέα τη άμυνα. Και τα τρία πιλωτικά αυτά προγράμματα ε, έκλεισαν επιτυχώ το πρώτο εξάμεινο του 2018. Με αυτές τις τρεις ερευνητικές ε, δραστηριότητες, το πιλωτικό πρόγραμμα έδωσε την δυνατική, τη πραγματική δυνατότητα να δούμε τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς μπορούν να συνεργαστούν με τον κλάδο, τον αμυντικό και με διάφορα ερευνητικά Ινστιτούτα. Ε, η υποεπιτροπή σας επίσης ε, βοήθησε στην πρώτη φάση του πιλωτικού και έδωσε τον πρώτο μορφότυπο για δραστηριότητες που συνεχεία αναπτύχθηκαν ανάλογα με το θέμα, την κατεύθυνση του project, παρακολούθηση του project ε, και τη κοινοβρασία που κέρδισε το διαγωνισμό. Το πιλωτικό πρόγραμμα ήταν σημαντικό γιατί για πρώτη φορά ελέγξαμε τι ε, συνθήκε για την έρευνα στον τομέα τη άμυνα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ετοίμασε το δρόμο για την ε, δρομολόγηση τη προπαρασκευαστική δράση ε, το 2017 για την έρευνα στον τομέα της Άμυνα. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι η διαχείριση των ε, project από τον οργανισμό μας ξεπερνάει τον τομέα της ε, έρευνας στο μη σκέλος, γιατί είμαστε επιφορτισμένοι για να εξασφαλίσουμε τη συνέπεια ανάμεσα στις, ε, σε αυτά που φτιάχνουν οι ανάδοχοι των έργων και για να κολλάνε αυτά τα πράγματα που αναπτύσσουν αυτοί με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες των κρατών μελών και τα υπουργεία, τις, ανάγκες των πραγματικές ανάγκες των Υπουργείων Άμυνας. Αυτό το πιλωτικό project έδωσε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε τομείς ε, που είχαν εντοπιστεί εκ των προτέρων. Συνολικά, Κάναμε μια αξιολόγηση ε, η οποία είναι πάρα πολύ θετική. Η συνεργασία με την Κομισιόν ήταν θαυμάσια και οι εκθέσεις από τους ανεξάρτητους παρατηρητές επίσης ήταν πάρα πολύ θετικές. Ε, θα ήθελα όμως να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες στα πιλωτικά προγράμματα, για τα πιλωτικά προγράμματα. Καταρχάς, η συνάδελφος μίλησε για αυτό το scoping paper της προπαρασκευαστικής δράσης και το πιλωτικό πρότυπο, ε, project εντάσσεται εκεί. Εδώ βλέπετε το βαθμό στον οποίο το project για το οποίο θα σας μιλήσω ε, εντάσσεται, που εντάσσεται, σε ποιο στρατηγικό κλάστερ επικοινωνίες, ε, intelligence, ε, πληροφορική, ε, αναγνώριση. Βλέπετε επίσης και τους τομείς τεχνολογίας και καινοτομίας που αντιστοιχούν. Λοιπόν, για να δείτε την ποικιλομορφία των project που καλύπτονται, ε, επέλεξα ένα project ευρώ μήνος και άλλα δύο για να σας μιλήσω <laughs> με λεπτομέρειες. Ε, για το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα ε, μιλάμε για μια δράση που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 434.000 ευρώ για 15 μήνες και 3 μήνες παράταση. Το project ε, ήταν επικεφαλής ε, ένα ακαδημαϊκός οργανισμός και τέσσερα κράτη-μέλη με νέες τεχνικές για προσαρμοσμένες ε, ουσιαστικές επιχειρήσεις ε, των συστημάτων και προτάθηκαν κάποιες λύσεις ε, με κάποια πειράματα που έγιναν σε μικρή κλίμακα, περιορισμένος ο προϋπολογισμός. Το να κλείσει αυτό το project με προσωμιώσεις, ε, θετικές κτλ. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξοδέψουμε τα λίγα λεφτά που έχουμε. Λοιπόν, σκεφτείτε ένα σενάριο όπου έχουμε ένα στρατόπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ξένη, όχι κατά ανάγκη φιλική μας χώρα. Έχουμε ένα μικρό ανεπάνδρωτο σύστημα το οποίο περίπταται πάνω από το στρατόπεδο για να εντοπίσει τις απειλές. Σε περίπτωση που υπάρχουν απειλές, ε, έχουμε μικρά ας πούμε ελικόπτερα ανεπάνδρωτα, τα οποία επιτίθενται κατά της απειλής. Αν χρειάζεται περαιτέρω επιθεώρηση, τότε θα έχουμε και ε, ανεπάνδρωτα συστήματα εδάφους. Όλα αυτά τα συστήματα, τα ανεπάνδρωτα, ε, συντονίζονται μέσω ενός συστήματος πληροφορικής. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε περισσότερες απειλές, ε, χρησιμοποιώντας όλους τους ε, drones που έχουμε στη διάθεσή μας. Εν συνεχεία, ε, συζητάμε τις δραστηριότητες που θα αναπτύξουμε μετά από τον εντοπισμό της απειλής, με το συντονισμό και συμμετοχή των Υπουργείων Άμυνα στο project αυτό. Αυτό δείχνει ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αμυντικές τεχνολογίες εν συνεχεία, ούτω ώστε να, τα να τις εντάξουμε σε αμυντικά προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν συνεχεία τα Υπουργεία Άμυνας των κρατών μελών. Προχωρώ στο πρόγραμμα ε, Οκεανή 2020. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο ε, ε, έγινε και, έγιναν και επιδείξει σχετικά. 36 ε, μήνες, 35,5 εκατομμύρια. Το, η κοινοπραξία ήταν από 15 διαφορετικά κράτη-μέλη με 42 φορείς ε, και συμμετείχε και ένας διεθνής οργανισμός. Ανοιχτή συνεργασία για ε, εποπτικές επιχειρήσεις στη θάλασσα με διάφορα συστήματα ανεπάντρωτα, αέρος, ε, θαλάσσης, υποθαλάσσια κτλ έχει, έγιναν πάρα πολλές επιδείξεις ε, στην Βαλτική και στη Μεσόγειο για να βρούμε καινοτόμε λύσεις για συγχώνευση ε, και χρησιμοποίηση από κοινού πολλαπλών πηγών ε, μαζί με συστήματα μάχης σε ένα ασφαλές δίκτυο, ούτω ώστε να έχουμε μία αναγνωρίσιμη θαλάσσια εικόνα. Το πρόγραμμα Οκεανή 2020 είναι ένα τεράστιο project με σενάρια σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο από ό,τι παλιότερα. Ε, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία ανάμεσα στα ανεπάντρωτα συστήματα. Είχαμε επιδείξεις με πολεμικά πλοία από διαφορετικά κράτη-μέλη, ε, προσγείωση επίσης των ανεπάντρωτων συστημάτων ε, σε πολεμικά πλοία. Έγιναν 7 μεγάλες συνεδριάσεις με θετικά συμπεράσματα για αυτό το πρόγραμμα. Η οργάνωση των πρώτων επιδείξεων ξεκίνησε και θα λάβει χώρα η, τα γυμνάσια αυτά, οι επιδείξει αυτές, στη Μεσόγειο ε, τον Οκτώβριο του 2019. Μεταξύ των συστημάτων για στρατιώτες έχουμε ένα άλλο project, Gross Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 1,5 εκατομμύρια ευρώ για 22 μήνες. Το, προς, ε, το project αυτό. Ε, ε, συμμετέχουν 7 κράτη-μέλη ε, και 9 εταιρείε. Θέλουμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα για προστασία στρατιωτών με πληροφορική, επικοινωνία, data, λογισμικό, αισθητήρε, sensors δηλαδή κτλ. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε κυρίως για τον εξοπλισμό σε λεπτομέρειες. Το βασικό είναι η διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, ε, οι οποίες συμμορφούνται με αυτή την αρχιτεκτονική δομή, καλό είναι να συνεργάζονται μεταξύ τους, να υπάρχει απαραίτητη επιμελητία για τις επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούνται. Έχουμε μια τυποποιημένη σύσταση του ΝΑΤΟ που θα χρησιμοποιήσουμε για την αρχιτεκτονική, ούτως ώστε να συμπληρώνουμε τις νατοικές δράσεις από ευρωπαϊκής Πλευρά και όχι να το ανταγωνιζόμαστε το ΝΑΤΟ. Ε, έχουμε γίνει, έχουν γίνει μελέτες ε, στον οργανισμό μου προηγουμένως ε, για να δούμε ποιες θα είναι οι τεχνικές προϋποθέσεις για το project. Είναι βασικό να αξιοποιήσουμε τα, κονδύλια που έχουμε τώρα, μέχρι τώρα τα πανίσει και το βασικό είναι να χρηματοδοτήσουμε κάποια project που θα οδηγήσουν σε νέες δραστηριότητες. Όπως αποδείχτηκε σε ένα εργαστήριο πρόσφατα με εμπειρογνώμονες, το project ε, έχει προχωρήσει και θα δώσει τα αποτέλεσματα που περιμένουμε, πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κράτη-μέλη, καθώς και οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ. Περνάω τώρα σε κάποια διδάγματα σχετικά με αυτές τις προπαρασκευαστικές δράσεις της Πάντερ και να σας δώσω κάποια παραδείγματα υλοποίησης. Δοκιμάζοντας ε, την συνεργασία μεταξύ της Κομισιόν και του Οργανισμού Αμήνης, έχουμε κάποιες διευθετήσεις, ε, κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και ε, υποβάλλουμε σε δοκιμές και ειδικέ εκθέσεις το οποίο είναι σημαντικό για το ρυθμιστικό πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων που θα πρέπει να έχει μια ισορροπία μεταξύ εγγυήσεων και επαρκούς ροής πληροφοριών, όπως και επαρκούς χρηματοδότησης, ώστε τα Υπουργεία Μήνης, που είναι οι τελικοί χρήστες, να έχουν ε, ε, επαρκή δικαιώματα πρόσβασης. Επίσης έχουμε ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερουμένους ε, φορείς για τον καλύτερο καθορισμό των θεματικών και λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαίτερες ανάγκες στον αμυντικό τομέα γιατί σε αντίθεση με την ε, έρευνα στον πολιτικό τομέα πρέπει να μένουμε στις θεματικές και να έχουμε και δράσεις παρακολούθησης λόγω της τεχνολογικής δυσκολίας στο πεδίο της άμυνας. Για τον οργανισμό αμήνης, τα διδάγματα δείχνουν ότι έχουμε δραστηριότητες και downstream και upstream. Για τους διαγωνισμούς των προπαρασκευαστικών δράσεων έχουμε δει ότι ο οργανισμός είναι απολύτως έτοιμος να αναλάβει το ρόλο της υλοποίησης και ήδη οικοδομούμε επί των διδαγμάτων, οικοδομώντας περαιτέρω τις ε, βέλτιστες πρακτικές που θα χρειαστούμε για τις μελλοντικέ ευρύτερης κλίμακας πάντερ. Η Κομισιόν συμφωνεί με, την με τη γενική αξιολόγηση και τις γενικές στοχεύσεις των προπαρασκευαστικών αυτών δράσεων και ότι έχουν καλύψει τους στόχους τους θα πρέπει βεβαίως να οικοδομήσουμε την απαλήτητη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών στον τομέα της άμυνας. Για τον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα των δράσεων αυτών, τα δύο πρώτα προγράμματα εργασία έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς και ήδη αναφέρθηκα στη δουλειά που μένει ακόμα να γίνει εκεί. Για τα κατάντι, γνωστά και ως downstream, Αυτό είναι ένα στοιχείο που χρειαζόμαστε προκειμένου να εκμεταλλευτούμε καλύτερα σε ένα πλαίσιο ενωσιακής χρηματοδότησης τα προγράμματα αυτά. Η απορρόφηση από τα κράτη-μέλη των συμπερασμάτων της έρευνας αυτής θα είναι η τελική δοκιμασία της επιτυχίας τους και αυτό μπορεί να γίνει με έργα παρακολούθησης εντός του Ταμείου του Αμυντικού και εντός εθνικών ή πολυεθνικών έργων ερεύνης, ώστε να αναπτύξουμε μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες. Και προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δράσεων, τα Υπουργεία Αμήνης θα έχουν κάποιες εναλλακτικέ για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, ό,τι και να επιλέξουν, ο Οργανισμός Αμήνης θα προωθεί στη συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων, αλλά βέβαια το πλαίσιο της υλοποίηση θα μείνει στα κράτη-μέλη. Για τα ανάντι τώρα. Ο ρόλος στην υποστήριξη των κρατών μελών είναι ο βασικός άξονας των πάντερ, των προπαρασκευαστικών δράσεων, με συναντήσεις συντονισμού, διαβούλευση στα κράτη-μέλη, αξιολόγηση των θεμάτων που έχουν υποβληθεί από τα κράτη-μέλη, το clustering και η καλύτερη επιλογή των υποθεμάτων. Και όλα αυτά προς την κατεύθυνση του μελλοντικού αμυντικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως εντός της όσρα που είναι το γενικό στρατηγικό θεματολόγιο θα πρέπει να αναπτύξουμε τα μελλοντικά προγράμματα υπό το Ταμείο Αμήνης και το βασικό αυτό θεματολόγιο όσρα ε, συνδυάζει μάλλον μια προσέγγιση top-down και bottom-up, συνδυάζοντας νέες τεχνολογίες και δυναμικό, ώστε να εναρμονίζονται καλύτερα οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες ε, αμήνης και η καλύτερη χρηματοδότηση των έργων. Ο ρόλος upstream του οργανισμού εξασφαλίζει ότι όλα αυτά θα πρέπει να συνδέονται και με τις στρατιωτικές αμυντικέ ανάγκε των κρατών μελών, γιατί η αμυντική έρευνα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι τεχνικέ προποθέσει θα καλύπτουν μελλοντικέ αμυντικέ ανάγκε, έτσι όπω αυτέ θα έχουν καθοριστεί από τα κράτη-μέλη. Συνολικά θα μπορούσα να πω ότι ο οργανισμό έχει διαδραματίσει και διαρματίζει και upstream και downstream έναν επιτυχή ρόλο στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και επιπροσθέτως οι δράσει αυτές δείχνουν ότι το θεσμικό αυτό πλαίσιο, ο διακανονισμός, είναι επιτυχής και αποτελεσματικός. Και υπάρχει αμοιβαία συνεργασία της Κομισιόν και του οργανισμού, ώστε η χρηματοδότηση των έργων αυτών να είναι επιτυχής και στο μέλλον. Με την κοινή εμπειρογνωμοσύνη του οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από διάφορους τομείς της αγοράς και της τεχνολογίας δίνει περισσότερα εχέγγυα για την τελική επιτυχία των έργων αυτών. Συμπερασματικά τα πιλωτικά αυτά έργα είναι πολύ χρήσιμες, πολύτιμες δοκιμές, τεστ για τη μελλοντική χρηματοδότηση. Υπό την οπτική γωνία των αναγκών της αμήνης, για την υλοποίηση που θα πρέπει να υπάρχει σε όλους τους ρόλους και σε όλη την αλυσίδα υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, ανάντι και κατάντι όπω λέγαμε. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ζητούσα τώρα από τους συντονιστές να τοποθετηθούν, ξεκινώντας τον κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ και για τις δύο παρουσιάσεις να συμπεράνω ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία στο μεταξύ έχουν συνηθίσει τόσο πολύ ο ένας τον άλλον ώστε να μην ε, υπάρχει πρόβλημα και να μην κάνει καμία διαφορά που δεν είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά των κρατών μελών. Έχετε συνηθίσει ο ένας τον άλλον, είστε εντάξει τώρα και ε, σε ό,τι αφορά τα έργα και τις ιδέες. Θα με ενδιέφερε να μάθω τελικά πώς τα επιλέξατε. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ε, είχε κάνει κάποια πιο προεργασία ή τα κράτη-μέλη σας επηρέασαν, σας έσπρωξαν προς τη μία την άλλη κατεύθυνση για την επιλογή των έργων υπήρχαν στρατηγικά έγγραφα, είτε είναι αυτή η παγκόσμια στρατηγική της Ένωσης ή ε, κάποιοι ειδικοί στόχοι. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στο Κοινοβούλιο, ε, πέρα από τον έλεγχο των οικονομικών ε, του πιλωτικού προγράμματος και των προσχεστικών δράσεων, ε, είναι ακριβώς αυτό ίσως να ρωτήσω και τους συναδέλφους ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εσείς πώς το βλέπετε. Και τα ερευνητικά αποτελέσματα ε, του πιλωτικού προγράμματος. Τι έγιναν. Συνεχίστηκαν με συνεργατικά προγράμματα. 1,5 εκατομμύριο δεν είναι πολλά χρήματα. Ε, κάπου, σε κάποιο αποτέλεσμα καταλήγεις. Μετά τι συνέχεια δίνεται. Άλλη ερώτηση. Όταν άρχισε το πιλωτικό πρόγραμμα, ε, τέθη ένα ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Λύθηκε αυτό το θέμα, τα συμφωνήσατε. Και με αυτό που έχετε πλέον αναπτύξει. Έκλεισε κανένα έλλειμμα ε, στους ε, μεγάλους στόχους, τους headline goals που είχαμε θέσει. Και για το μέλλον τώρα, ε, για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, τι θα γίνει με το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης. Γιατί πρόκειται για μεγαλύτερα ποσά, μήπως χρειάζεται πιο πολύ κόσμο. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις και παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα κάπως και έτσι έχασα το πρώτο τμήμα των παρουσιάσεων. Ίσως να αναφερθήκατε ήδη δηλαδή σε αυτά που θέλω να πω. Η δική μου κύρια ανησυχία και της ομάδας των Πρασίνων και νομίζω και σημαντική ανησυχία και της κοινωνίας των πολιτών είναι η διαφάνεια και μια αποτροπή της συγκρούσεως συμφερόντων. Υπάρχει το εξή πρόβλημα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα πράγματα για το έργο της ομάδος των προσωπικότητων που συμβουλεύουν την Κομισιόν. Τα θεματολόγια, οι διατάξεις θα είναι δημόσια διαθέσιμα. Πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι θα συμβαίνει στην ομάδα αυτή. Επίσης, εξ όσων γνωρίζω, έξι από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ομάδα τη συμβολευτική αυτή είχαν συμμετάσχει σε διαφορετικούς διαγωνισμούς των πάντερ. Δεν είναι αυτό σύγκρουση συμφέροντος. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε ήδη, αλλά αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ, η κυρία Λόζινγκ. <coughs> Ευχαριστώ πολύ. Η δική μου ερώτηση έρχεται να επαναλάβει λίγο την ερώτηση της κυρίας Βαλέρο. Σε μερικά σημεία θα μπορούσα ίσως να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Οκεανή 2020, 35 εκατομμύρια με διαφορά το μεγαλύτερο έργο της προπαρασκευαστικής δράσης. Διαβάζω τον κατάλογο των συμμετεχόντων και των επωφελουμένων εταιριών εμπολής. Και τι διαπιστώνω, σχεδόν όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ομάδα υψηλού επίπεδου που έκανε έκθεση το 2016 το Φεβρουάριο και ε, ζήτησαν αμυντικό ε, οργανισμό συμμετέχουν τώρα Λεωνάρδο, ΣΑΠ, Ίντρα, MDA και πάει λέγοντα. Όλοι αυτοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα για του ωκεανού. Και αν το τραβήξω λίγο, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανεί. Η βιομηχανία έγραψε μόνη της το πρόγραμμα αυτό που θα την ενισχύσει. Και τι γίνεται με τη σύγκρουση συμφερόντων, ιδιαίτερα σε τόσο προβεβλημένες εταιρείες. Πώς μπορεί αυτή να αποφευθεί υπήρχαν και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ε, που μπορεί κανείς να αποδείξει ότι δεν έχουν σχέση με την αμυντική βιομηχανία εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους οποίους να ανατέθηκε ο έλεγχος ε, των αιτήσεων. Ας πούμε, το έργο του 2020 για τους ωκεανούς, παραθέτω, παρακολούθηση των ωκεανών και παρεμπόδιση ε, και παρακολούθηση παρεμπόδισης ναυσιπλοείας και θαλάσσιας κυκλοφορίας. Πολύ θολά αυτά και συγκεχημένα. Για ποιο λόγο. Τι έργο είναι αυτό για την καταπολέμηση της μετανάστευσης, μήπως. Ή... Και αν ναι, γιατί συγκεκριμένα και πώς θα το κάνετε αυτό. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Και προς τους δύο ομιλητές. Τώρα, μετά από τα χρόνια που έχουμε παρέλθει, πώς αξιολογείτε την συνεισφορά και των πιλωτικών έργων και των προπαρασκευαστικών δράσεων για την οικοδόμηση δικτύων. Επίση, ε, πώς αξιολογείται την ποσόστοση των περιφερειών και των χωρών στην συνεισφορά αυτή. Γιατί συζητώντας στην Επιτροπή το, τα επίπεδα συμμετοχής Εξεπλάγην όταν άκουσα ότι εντός μίας και μόνης χώρας, μιας από τις πιο προηγμένες όπως η Γερμανία, υπήρξε πολύ μεγάλη απόκληση μεταξύ των ανατολικών και δυτικών περιφερειών της χώρας στην συνεργασία αυτή. Έχετε σημειώσει κάποια βελτίωση ή πιο εκπεφρασμένη βούληση συμμετοχής και σε διασυνοριακά έργα, αντίστοιχα. Ποιος θεωρείται ότι θα είναι ο καλύτερος μελλοντικός τρόπος συνεργασίας, αντιστοίχως βεβαίως προς το πώς θα πάνε τα πράγματα στο Brexit. αλλά θεωρώ ότι η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο ούτως ή άλλως είναι ύψης της σημασίας, γιατί η συνεισφορά της χώρας αυτής στα θέματα ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντική. Τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει, να προβλέψει. Και βεβαίως σε επίπεδο του οργανισμού το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παρόν, αλλά δεν είμαι απόλυτα βέβαιη πώς αυτός ο κόμβος μεταξύ του οργανισμού EDA και της Κομισιόν θα λειτουργήσει για την Ευρώπη μετά το Brexit. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ίσως κάποια περαιτέρω σχόλια τεχνολογικών προβολών, προβλέψεων σχετικά με το ποιο ήταν το σημείο εκκίνησης και ποιο περιμένουμε να είναι το τελικό αποτέλεσμα των διαγωνισμών των τεχνολογικών και τι φύσεως έργα περιμένουμε να έχουμε. Δηλαδή περισσότερο θα έχουμε έργα θεωρητικής ανάλυσης, brainstorming ή πρακτικής χρησιμότητος σε υφιστάμενα πεδία. Νομίζω ότι και από την αίθουσα και από την έδρα αυτές είναι οι ερωτήσεις, άρα με την ίδια σειρά, αν θέλετε παρακαλώ, απαντήστε στις διαφημιστικές αυτές ερωτήσεις. Κυρία μου, εσείς πρώτα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να απαντήσω πρώτα σε ερωτήσει του κυρίου Γκάλερ πόθεν ε, τα έργα και σε τι βασιστήκαμε για να τα επιλέξουμε. Το εξήγησα προηγουμένως. Συστήσαμε ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία εξέτασε την προπαρασκευαστική δράση. Η προπαρασκευαστική δράση δεν είναι νομοθέτημα, προέρχεται από το δημοσιονομικό κανονισμό. Οπότε δεν μπορούμε να συστήσουμε επιτροπή κανονικά που να παρτίζεται από τα κράτη-μέλη. Και ε, συγκαλέσαμε λοιπόν μια ομάδα πυρογνωμόνων που λειτουργεί αντίστοιχα με τις ομάδες των κρατών μελών και προετοιμάζει το ετήσιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αμήνης, το εξήγησα και αυτό εισαγωγικά, είναι παρατηρητής εκεί. Upstream input, ε, και κάνει προτάσεις με βάση τις διαδικασίες ή τα σχέδια που υπάρχουν ήδη ε, προτεραιότητες ε, στα πλαίσια ε, των δυνατοτήτων, των ικανονίτων και του δυναμικού που χρειάζονται. Εκεί βασιστήκαμε. Αυτό είναι το upstream που λέγαμε το ανάντι. Αλλά και τα κράτη-μέλη κάνουν τις προτάσεις τους πέρα από την ομάδα αυτή των εμπειρογνωμόνων. Δεν ακολουθήσαμε ένα προς ένα τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης ή ε, το δικό του έτσι, προγραμματισμό. Συνεννοηθήκαμε και με τα κράτη-μέλη που έχουν τις προτεραιότητές τους και τις κατέθεσαν. Ε, σε αυτή τη βάση λοιπόν βγήκε το πρόγραμμα εργασίας τα κείμενα της προκήρυξης των διαγωνισμών, αυτά καθ' αυτά, ε, προέκυψαν μετά από συνεννόηση με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσανατολίστηκε ε, στη πραγματογνωμοσύνη που υπάρχει στα κράτη-μέλη και τα εμπιστεύτηκε γι' αυτό. Για τον έλεγχο του προϋπολογισμού, πώς έγινε αυτό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αμήνης δουλεύει όπως κάθε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εντός των δημοσιονομικών κανόνων, απολύτως. Ρωτήσατε ειδικά ε, τι γίνεται με το λογιστικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης, αν το αναγνωρίζουμε. Μα όπως και κάθε οργανισμός έχει τις διαδικασίες. Έχει ένα εσωτερικό λογιστικό έλεγχο πρώτα, για να αξιολογήσει τι γίνεται με την εκτέλεση ε, των έργων και των προπαρασκευαστικών δράσεων και αν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες δομές, μηχανισμοί, κανόνες κτλ. Και αυτό μελετήθηκε και εξετάστηκε ε, σχολαστικά. Πώς έγινε η συνεργασία και τα υπόλοιπα θα τα αφήσω να απαντήσει ε, ο κύριος Τιλμπιργκερ αν συνηθίσαμε να συνεργαζόμαστε ε, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μήνης. Ε, κοιτάξτε, δεν είναι το ίδιο πράγμα να είσαι θεσμικό όργανο της Ένωσης, βλέπει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συνεργάζεσαι με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μήνας, που είναι διακυβερνητικό όργανο και οργανισμός των κρατών μελών. Οι δομές είναι διαφορετικές βεβαίως, οπότε και χρειάζεται και στην πρακτική εφαρμογή κάποια συζήτηση ε, για να συνεννοηθούμε και να καταλήγουμε κάθε φορά. Ε, αυτό λειτουργήσε πάντως στα πλαίσια ε, των προπαρασκευαστικών δράσεων για την άμυνα. Αλλά υπάρχουν διαφορές στη διακυβέρνηση. Και ως προς τις διαδικασίες και ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι διαφορετικός. Αυτό το αναγνωρίζουμε, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Στην πράξη, στην εφαρμογή και την υλοποίηση όλων αυτών, στα πλαίσια της συμφωνίας ανάθεσης ε, λειτουργήσαμε πάρα πολύ καλά και ήταν αγαστή η συνεργασία. Μια που μιλάω γερμανικά, να απαντήσω και στην κυρία Λόζινγκ στα γερμανικά. Η συνεργασία για τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράση. Σας παρακαλώ να μην γίνεται σύγχυση με το GOP, Group of Personalities, την ομάδα προσωπικότητων και την επιλογή των θεμάτων ή των έργων στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής δράσης. Υπάρχει μια ομάδα προσωπικότητων που έχει ένα πάρα πολύ ειδικό ρόλο. Ε, ήταν παρούσα σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο έτσι ώστε να απευθύνει συστάσεις. Πώς μπορεί μια κοινή έρευνα και κοινά ερευνητικά προγράμματα στην άμυνα να ε, διεξαχθούν στην Ένωση. Αυτές οι συστάσεις στη συνέχεια ε, έδωσαν μια έκθεση και εκεί τελειώνει η ομάδα προσωπικότητων και ο ρόλος της. Ε, δεν είχαν κανένα τρόπο να επηρεάσουν την επιλογή των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αυτό όπως και στην έρευνα για πολιτικούς σκοπούς, η επιλογή και η αξιολόγηση των ε, έργων ε, γίνεται μετά από τις ε, προτάσεις που υποβάλλουν ερευνητικά Ινστιτούτα, κοινοπραξίες, επιχειρηματικοί όμιλοι, πανεπιστήμια, όποιος θέλει να συμμετάσχει εκεί. Αυτά τα αξιολογούν και τα επιλέγουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και αυτά τα εξήγησα προηγουμένως και επιλέγονται στα πλαίσια ε, ε, μιας ε, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έτσι ονομάζεται. Και υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να επιλεγούν. Χρειαζόμαστε μια ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε συγκεκριμένους τομείς όπου χρειάζεται να γίνει και το ερευνητικό πρόγραμμα. Άρα να υπάρχει τεχνική και τεχνολογική γνώση για να μπορέσουν να τα αξιολογήσουν. Και όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες έρχονται ως πρόσωπα, ad personam, σε προσωπική βάση, δεν εκπροσωπούν κανέναν, θα πρέπει να έχουν ειδική έγκριση ε, και άδεια για πρόσβαση σε ε, διαβαθμισμένα έγγραφα και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες που ε, προσκαλούνται να αξιολογήσουν ένα έργο και το ίδιο έργο, το έργο αυτό. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση η ομάδα προσωπικότητων, αυτό το group of personalities με τους εμπειρογνώμονες που επιλέγουν τα προγράμματα. Και τελευταίο, για να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Βαλέρο, αλλά νομίζω σχεδόν την απάντησα ήδη ε, για την ομάδα των προσωπικότητων, GOP. Ε, για το εάν δημοσιεύουμε τα πρακτικά και τις ημερήσεις διατάξεις, είναι και απόφαση της διαμεσολαβήτριας αυτή, πώς να το πω Μιλήσατε για διαφάνεια. Ο τρόπος που χειρίζεται τη διαφάνεια ομάδα προσωπικότητων δεν έχει να κάνει με ε, έλλειψη επαγγελματισμού ή ε, λαθροχειρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτή η ομάδα δεν ήταν τυπικά και επίσημα ομάδα εμπειρογνωμόνων και δεν μας δέσμευαν όλες αυτές οι δεσμεύσεις νομικές που έχουμε για τις ημερήσεις διατάξεις των ομάδων εργασίας ή τα πρακτικά, διότι δεν εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Ταυτόχρονα όμως είπε η διαμεσολαβήτρια ότι ήταν αυτή μια συμβουλευτική επιτροπή η οποία έκανε συστάσεις στην Επίτροπο Μπιανκόσκα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και ενώ δεν υπάρχει μεν υποχρέωση ε, να δημοσιεύονται αυτά τα έγγραφα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καλό θα ήταν να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε η Δεμεσολαβήτρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις για το πώς προτίθεται να το κάνει και θα την καταθέσουμε αυτή την πρόταση. Ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί, δεν θέλω να σας αποκαλύψω τώρα πότε θα γίνει και πώς ακόμα ε, αναμένεται η έγκριση από την ιεραρχία μας. Αυτή τη στιγμή όμως ε, δημοσιευθεί αυτό και εγκριθεί από τη διαμεσολαβήτρια θα σας ε, ενημερώσουμε και θα διαθέσουμε και θα δημοσιεύσουμε τα απαραίτητα έγγραφα. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αλλά πρώτα ο κύριος Μετά την τοποθέτηση του ομιλητή μας θα δώσω το λόγο στους βουλευτές για ερωτήσεις, αλλά υπάρχει και θέμα χρόνου προσοχή λοιπόν. Να απαντήσω πρώτα σε ερωτήσεις του κυρίου Γκάλερ. Ε, πολλά απαντήθηκαν από την κυρία Κάιντς Χούμπερ. Η επιλογή των προγραμμάτων και των έργων είναι από κάτω προς τα πάνω. Ε, τα κράτη-μέλη και σε συνεργασία μεταξύ τους ε, κουβέντιασαν ποιες είναι οι σημαντικές υποχρεώσεις που είχαμε και στο πιλωτικό πρόγραμμα και στην προπαρασκευαστική δράση. Και στο μέλλον αυτό θα πρέπει να είναι διαφορετικό. Πρέπει να δούμε γενικά την έρευνα που χρειάζεται για την άμυνα. Γιατί στην αρχή αυτό που μας ενδιέφερε περισσότερο ήταν η συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης και λιγότερο ποια είναι τα συγκεκριμένα έργα που θα επιλεγούν, γιατί ήταν περιορισμένη η χρηματοδότηση, τα ποσά δηλαδή. Βεβαίως επιλέξαμε τα σημαντικά έργα, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι τομείς που μας ενδιαφέρουν για την έρευνα, την αμυντική. Σε σχέση με τους οικονομικούς πόρους και την προοπτική τους, Στη Συμφωνία Ανάθεσης ορίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβανομένη στη ΣΟΛΑΦ και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί ανα πάσα στιγμή να ελέγξει μέχρι και μία πενταετία ε, μετά την ολοκλήρωση του έργου ε, τα οικονομικά του συγκεκριμένου έργου. Δηλαδή έχει τον έλεγχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί ήδη ανα πάσα στιγμή να εξασφαλίσει ε, τα όσα ισχύουν και για τον εαυτό τη. Ό,τι ισχύει για τα προγράμματα της Κομισιόν ισχύει και για μας. Και όπως σας είπα, στο πιλωτικό πρόγραμμα δόθηκε συνέχεια. Υπήρξε μια τέτοια πρωτοβουλία. Το Euroswarm, αυτό το ευρωσμήνος, αυτό είναι κλασικό στην έρευνα. Ορισμένοι ενδιαφέρονται αμέσως ε, να πούν τι συνέχεια θα δώσουν και πώς θα μεταφραστεί το αποτέλεσμα της έρευνας στην πράξη και άλλοι είναι πιο διστακτικοί. Έκλεισαν ελλείμματα και κενά γιατί επιλέγησαν έτσι τα, τα προγράμματα που να οθήσουν τα κράτη-μέλη να εκφράσουν ενδιαφέρον. Και για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο που θα έχει περισσότερη χρηματοδότηση χρειάζεται φυσικά και περισσότερο προσωπικό. Αν και ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας έχουμε διαχειριστεί προγράμματα ε, της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ε, που χρηματοδοτήθηκαν τα κράτη-μέλη. Ήταν από χρηματοδότηση εθνική, τώρα είναι για ενωσιακή χρηματοδότηση. Για την κυρία Λότζιν να προσθέσω κι εγώ κάτι, αν μου επιτρέπετε. η επιλογή των θεμάτων δεν έγινε από την ομάδα προσωπικότητων, αλλά με πρόταση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εκεί αποφασίστηκε ποια είναι τα θέματα που θα μπουν στο πρόγραμμα εργασίας και στην προκήρυξη διαγωνισμών. Και ε, εκεί επιλέξαμε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, με βάση βεβαίως τι γνώσεις τους και την πραγματογνωμοσύνη, αλλά δεν επιτρεπόταν να έχουν και σύγκρουση συμφερόντων. Αν ανήκαν σε κάποια εταιρεία που συμμετείχε σε μια προκήρυξη ή είχε έναν υπεργολάβο να συμμετέχει, προφανώς αποκλείοντο από την ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Δηλαδή, από τη μια έχουμε στρατηγική ε, προσφορά, ας πούμε, προτάσεις με την ομάδα προσωπικότητων, η οποία διαλύθηκε και στη συνέχεια ε, ε, είχαμε υποβολή ε, ανταγωνιστική διαφόρων ομίλων και κοινοπραξιών για τα έργα. Και υπήρχαν και μεγάλες εταιρείες και μεγάλοι όμιλοι οι οποίοι χάσανε και δεν επελέγησαν. Ήταν πραγματικά ανεξάρτητοι, σας διαβεβαιώ, το ελέγξαμε και προσωρινά είχαμε και κάποια ονόματα ε, όπου αργότερα είδαμε ότι υπάρχει μια πρόταση, ε, μια υποβολή αίτησης ε, που συνδέεται με το συγκεκριμένο πρόσωπο η εταιρεία και τον αποκλείσαμε από τον κατάλογο. Νομίζω να απάντησα και ελπίζω να απαντά και στην ερώτηση της κυρίας Βαλέρο. Μιλήσατε στα γερμανικά να πω κάτι για το συγκεχημένο που είπατε και το θολό και το αόριστο ε, για το πρόγραμμα Οκεανή 2020. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η πρόταση έχει γίνει αρκετά ευρεία, έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο για να έρθουν διάφορες προτάσεις από διάφορες κοινοπραξίες. Δηλαδή στην προκήρυξη θα πρέπει να είναι αρκετά γενικόλογη η διατύπωση για να έρθουν διάφορες προτάσεις και ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Δεν πρόκειται για τη μετανάστευση, ούτε για την ασφάλεια. Για την άμυνα πρόκειται, δηλαδή αμυντική έρευνα, στρατιωτική. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε ε, για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί και την αμυντική έρευνα που μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Και πρόκειται για σενάρια. Ας πούμε, έχουμε πολεμικά πλοία σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ εχθρικό ενδεχομένως να είναι σε θέση να ε, εξασφαλίζουν την άμυνά τους και να χρησιμοποιούν drones για να αποτυπώνουν την εικόνα από τον αέρα, να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, για να αποκαλύψουν κάποια απειλή και κάποιο κίνδυνο. Δεν είναι καθόλου έρευνα ασφαλεία για τη μετανάστευση και τη φύλαξη των συνόρων. Είναι κλασικές ναυτικές ε, δυνάμεις και αυτό, γι' αυτό δημιουργήθηκε και το πρόγραμμα Οκεανός 2020. Um, cross-border work together is, really uh, uh, incentivized. Έχουμε και την προπαρασκευαστική δράση και είδαμε τη σημασία της ε, στο Ωκεανός 2020 όπου συνεργάζονται 15 κράτη-μέλη. Ε, είναι εντυπωσιακό πόσοι φορείς συνεργάστηκαν, έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το μέγεθος του project ε, και την κοινοπραξία. 15 κρατη και 42 εταιρείες, φορείς συμμετείχαν σε αυτή την ε, κοινοπραξία. Ήταν μια διασυνοριακή συνεργασία και αυτή ακριβώς είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Τελευταίο ερώτημα, ε, το Tech4 είναι το Horizon Scanning το επιπλέον είναι ότι πρέπει να αποφασίσεις τι είδους ε, ερευνητικό πεδίο είναι σημαντικό για την ανάπτυξη δυνατοτήτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελικά για αμυντικούς σκοπούς. Πρέπει δηλαδή να εντοπίσεις θέματα τα οποία αξίζουν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τα κράτη-μέλη ή από άλλους πόρους. Ευχαριστώ. Πράγματι, ο κύριος Γκάλερ θα κάνει μια ερώτηση, αλλά πολύ σύντομα γιατί πρέπει να κλείσουμε αυτό το θέμα. Λιγότερο ερώτηση είναι και μάλλον επιβεβαίωση των λεχθέντων προηγουμένως. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη που κυκλοφορεί ότι ε, έγραψε μόνη της το πρόγραμμα η βιομηχανία. Αυτό απαντήθηκε και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2013 συμμετείχα και εγώ είχαμε μια έκθεση για ε, την ε, ευρωπαϊκή ε, βιομηχανική βάση για την άμυνα και εκεί ζητούσαμε την προπαρασκευαστική δράση. Ήδη από το 2013 το ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή έχουμε αναθέσει πολιτικά και εμείς και από το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει αυτό. Αργότερα το Συμβούλιο. Εξού και στον προπολογισμό του 2015 για πρώτη φορά ε, αποφασίσαμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η προϊστορία. Και δεν κατέβηκε η βιομηχανία να σχεδιάσει κανένα πρόγραμμα για να το ε, κόψει και να το ράψει στα μέτρα της ε, και για ίδια συμφέροντα. Μάλιστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τους δύο διακεκριμένους ομιλητές. Η υποεπιτροπή μας, η ΣΕΝΤΕ, πρέπει να συνεχίσει τη διερεύνηση αυτό το θέμα, αυτού του θέματος και οι ευρωβουλευτές ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Παρακαλώ, χειροκροτήστε τους ομιλητές μας μαζί μου. Θα περάσουμε αμέσως στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Μην βγείτε από την αίθουσα. Colleagues, please be seated. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Okay, now we can start. It uh, Αρχίζουμε. Με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω στη συνεδρίασή μας τον αναπληρωτή συμμαχικό διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στρατηγό Sir James Rupert Everard, γνωστό σε πολλούς από εσά. από το ΝΑΤΟ. Μέχρι το τέλος του περασμένου μήνα έπρεπε να επισκεφτούμε τη Μόντς. Αλλά ε, λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπόρεσα να πάω. Ο στρατηγός όμως δέχτηκε την πρόσκλησή μας σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω πραγματικά είχαμε καιρό να ανταλλάξουμε απόψεις με τον στρατηγό για την κοινή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, καθώς και για την εκτίμησή σας για τις απειλές στην ασφάλεια της Υπήρου μας. Έχετε το λόγο, στρατηγέ μου. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία απλή αφήγηση δύο λεπτών για να εξηγήσω τα τελευταία 74 χρόνια ιστορίας μας. Και το κάνω επίτηδες, ξέροντας ότι δεν υπάρχει ένα και μόνο αφήγημα στη Δύση, στη Ρωσία ή στα κράτη, ανάμεσα στις δύο αυτές δυνάμεις, ε, που εξηγούν την ε, σημερινή γεωπολιτική μας κατάσταση. Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες Ε, για τις αιτίε της αστάθειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Το περισσότερο μισό του δεύτερου, για το περισσότερο από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, υπό την ε, στεναρή ηγεσία της ε, Αμερικής, τα κράτη, τα έθνη του ΝΑΤΟ ετοιμάστηκαν σε μεγάλο βαθμό και με μεγάλο τίμημα για ένα πόλεμο ο οποίος δεν έλαβε χώρα. Το να πολεμήσουν αυτό το μη πόλεμο θεωρήθηκε πολύ σημαντικό και στην συμμαχία και η άμυνα και η αποτροπή έγινε βασικό μέλημα, αν όχι το μόνο μέλημα των ενόπλων δυνάμεων. Φυσικά κερδίσαμε. Στο τέλος του ψυχρού πολέμου, ε, με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, γιορτάσαμε την παγκόσμια νίκη, το παγκόσμιο θρίαμβο της φιλελεύθερης δημοκρατίας και φανταστήκαμε μια νέα παγκόσμια τάξη όπου αναφέροντας τι είπε ο George W. Bush, τα έθνη του κόσμου, η Ανατολή και Δύση, ο Βορράς και ο Νότος μπορούν να ζήσουν με ευημερία και αρμονία. Αυτή τη σύντομη χρονική στιγμή άλλαξαν όμως οι προτεραιότητες και πολλά έθνη έσπευσαν να εξασφαλίσουν ένα μερίδιο της ειρήνης και οι ευρωπαϊκές αμυντικές ταπάνες έπεσαν κάθετα ε, από 20 έως 32% ανάλογα με τις ε, πηγές που χρησιμοποιείς ανάμεσα στο 1995 και στο 2015. Άλλαξε τότε λοιπόν ε, η εστίασή μας και απομακρυνθήκαμε από τη συλλογική άμυνα στις ε, ειρηνευτικές αποστολές, στις ε, εξαιρετικές αποστολές και επιχειρήσεις, στην αντιμετώπιση των εξεγέρσεων, οικοδόμηση δυναμικού και στην αντιμετώπιση τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού. Το 2014 λοιπόν με κατάπληξη είδαμε ότι η Ρωσία προσάρτησε την Κρυμαία και παρενέβη στην Ουκρανία, μία πράξη η οποία οδήγησε στην επιστροφή του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό άλλαξε άρδιν το περιβάλλον ασφαλείας ε, Ευρώπης, ε, των Ευρώπης και Ατλαντικού, Ευρωατλαντικής Συμμαχία, α πούμε και είμαστε έτοιμοι τώρα να αντιμετωπίσουμε φορείς οι οποίοι αμφισβητούν τη την ε, διεθνή τάξη αλλά δεν έχουμε την ετοιμότητα να επιστρέψουμε στη συλλογική άμυνα. Ακόμα και τώρα, και τότε και τώρα, αντιμετωπίζουμε όλα τα μεγάλα στρατηγικά σοκ και σεισμούς και μετασεισμούς του 21ου αιώνα, τις επιθέσεις της 11ης ε, Σεπτεμβρίου, ε, τη χρηματοπιστωτική κρίση το κράχ, τη μεταναστευτική κρίση, ε, την Αραβική Άνοιξη, την αντίληψη για την απεμπλοκή των ΗΠΑ από τις δημόσιες και διεθνείς υποθέσεις και προβλήματα και διαιρέσει στην Ευρώπη για τις αξίες της. Τώρα το ΝΑΤΟ αντιμετωπίσει τη Ρωσία που είναι ένα κράτος και ένα μη κρατικό καρκίνωμα την τρομοκρατία. Ε, και παρότι δεν είμαστε σε μια φάση στρατηγικής αντιπαράθεσης, είμαστε σε μια φάση στρατηγικού ανταγωνισμού. Τώρα ας πάμε στη Ρωσία. Μπορείτε να πείτε ότι η Ρωσία ε, είναι και πάντα ήταν κολλημένη ε, σε στρατηγικούς φραγμούς, ας πούμε το σιρού παραπέτασμα, ε, ζώνες επιρροής, ε, κοινωνικός έλεγχος, ούτως ώστε να προλάβει τις παρεμβάσεις στην καλύτερη περίπτωση ή τις επαναστάσεις στη χειρότερη. Ε, και μπορείτε να ταυτιστείτε με μια χώρα η οποία ε, πλήττεται, ταλανίζεται από φόβους ότι θα την καταλάβουν. Ε, η Ρωσία δεν είναι η αρκούδα στο λιβάδι ανησυχεί για τη θέση της στον κόσμο, μπορείτε να πείτε, και έχει μια αμυντική στρατηγική. Αλλά μπορείτε να πείτε βεβαίω ότι αντιμετωπίζουμε και μια πιο επικίνδυνη Ρωσία σήμερα. Μια Ρωσία η οποία είναι αποφασισμένη να ξαναεμφανιστεί ω υπερδύναμη και αν χρειαστεί και όταν χρειαστεί να δημιουργήσει πρόβλημα και να διασαλεύσει την ε, παγκόσμια τάξη που προέκυψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει έναν αμυντικό προπολογισμό η Ρωσία που θα πρέπει να τον κρίνεται όχι με βάση τα δολάρια που ξοδεύει, αλλά με βάση το ισοδύναμο αγοραστικής αξίας, άρα δεν είναι 67 δισεκατομμύρια αυτά που ξοδεύει, αλλά περίπου 200 δισεκατομμύρια αυτά που ξοδεύει η Ρωσία για την άμυνα. Η Ρωσία ε, επενδύει ε, για να αποσταθεροποιήσει τον ευρωατλαντικό χώρο όχι για να κερδίσει έναν ε, μακροσκελή πόλεμο, αλλά μέσω συνεχών εκστρατιών, ε, εκφοβισμού, με υβριδικές δραστηριότητες. Ο Λίνδι Φρέντς είπε ότι κάνει ένα συνεχή ε, πόλεμο, ε, χροπραξίες, με παραπληροφόρηση, αποσταθεροποίηση, παρα, διασαλεύσεις, απάτες και καταστροφή προφανώς χρησιμοποιεί αυτούς τους λεγόμενους βραχίβιους πολέμους με γρήγορες, ε, γρήγορα εκτελεσμένες ε, εκστρατείες, σαφείς γεωγραφικούς στόχους, 30 με 60 μέρες διάρκειας. Παράλληλα, βλέπουμε διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες, ε, οι οποίες προσπαθούν να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους και να επιτεθούν στις πόλεις μας, να προσπαθούν να εξασφαλίσουν προχωρημένα συμβατικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής, ούτως ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση του αγώνα τους. Για να περάσουν από την τάξη σε μια νέα τάξη, ε, οι Ρώσοι που τους αρέσει περισσότερο και οι τρομοκρατικές ομάδες σε μια νέα τάξη, ε, στην, από την αταξία σε μια νέα τάξη και τελικά στην ε, συνθηκολόγηση της δύση. Λοιπόν, ε, ο συμμαχικός διοικητής ε, στην Ευρώπη και η, γραμματεία του, Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ έχουμε μία, αναπτύξει μία ε, βασική στρατηγική για να, τις, να αντιμετωπίσουμε τις στρατηγικές προκλήσεις από το 2014 και ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές προκλήσεις. Θέλουμε αυτή η νέα στρατιωτική στρατηγική να ολοκληρωθεί. Τι περιμένω από αυτήν. Καταρχάς, αυτή η στρατηγική θα αποδειχθεί ε, αποτελεσματικό εργαλείο για να πετύχουμε μια συνεπή στρατιωτική στάση στις δραστηριότητε ε, που προωθούμε. Δεύτερον, να επιστρέψουμε σε μια πραγματική ετοιμότητα. Και τρίτον, μια και είμαστε συμμαχία, θα μπορέσουμε να δείξουμε την αντοχή μας, ε, να ανταγωνιστούμε συλλογικά, να ελέγξουμε το χώρο ασφαλεία μας, να μην δεχτούμε προκλήσεις και να δείξουμε ότι έχουμε ικανότητα για μακροσκελείς πολέμους και αν χρειάζεται να δείξουμε ότι η ανώτατη δύναμη της συμμαχίας να μπορεί να αντέξει σε, στο χώρο και στο χρόνο. Ε, ανέφερα τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει από το 2014. Ε, ε, θα ξέρετε ε, τι έχει συμβεί. Ε, υπάρχουν οι σύνοδοι κορυφή τη Βρυξέλλε, δεν θα τα καλύψω αυτά. Απλώ από το 2014 έχει μετασχηματιστεί η συμμαχία. Ε, επικεντρώνουμε ξανά στην αποτροπή. Πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο άμυνας και ασφάλειας ε, γίνεται πολύ πιο κατανοητό στο ΝΑΤΟ, αλλά και σε άλλους ε, χώρους και φόρουμ. Χάρη στις προσπάθειες Φεντερίκα Μουγκερίν για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι ε, και τι δεν είναι αυτή, αυτό το μοντέλο. Η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια είναι πολύ πιο περίπλοκη σήμερα και έχει συμπεριλαμβάνει κρατικού και μη κρατικού φορεί, τρομοκρατία, υβριδικέ απειλέ, κλιματική αλλαγή, οικονομική αστάθεια και έλλειψη ασφάλεια στην ενέργεια, στον ενεργικό αναφοδιασμό. Αναγνωρίζει ότι οι λύσει είναι και πολιτικέ αλλά και στρατιωτικέ και καταλαβαίνει τη σχέση μεταξύ τη άμυνα και τη ανάπτυξη μεταξύ της διαχείρισης των κρίσεων και της ε, συμφιλίωσης και ότι η επιτυχία αφορά, είναι και των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και η ενίσχυση όλων των εταίρων του ΝΑΤΟ ε, σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο κατανοητό σήμερα, όταν δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην επένδυση ε, στην στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και στη συνεργασία πιο στενά με βασικούς εταίρους, Αφρικανική Ένωση, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ και αυτή η διευθέτηση μπορεί να είναι να μας οδηγεί σε μία συμπληρωματικότητα και όχι ανταγωνισμό. Όχι στατικική αυτονομία ή συνεργασία, αλλά συνεργατική αυτονομία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρκετή δύναμη. Το Βερολίνο Plus είναι ένας μηχανισμός για αυτή την στρατηγική εταιρική σχέση Βερολί, ε, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ καλό. Το 2002 οι αρχιτέκτονες του Βερολίνου Plus σκέφτηκαν τα πράγματα ε, με κάθε λεπτομέρεια και σκέφτηκαν ε, ότι ένα ευρωπαϊκό ε, αρχηγείο που θα βασίζεται στο ΣΕΙΠ, το έχουμε ξεχάσει τώρα, θα έδινε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρόσβαση στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Ε, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ που δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο, στο μέλλον και να ε, έχουμε σαν σκοπό να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε το Βερολίνο Plus. Ε, Εκτό από αυτό, ε, η συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ βασίζεται γενικά σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του διεθνού προσωπικού του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 75 κοινέ προτάσει σε τομεί κοινού ενδιαφέροντο και στρατηγικό και επιχειρησιακό, ε, διαχείριση κρίσεων, υποστήριξη της διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας, καθώς και ανάπτυξη του αμυντικού δυναμικού. Ε, οι προσδοκίες μας είναι ότι αυτό σε πολιτικό επίπεδο ε, έχει θέσει τους, τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας άλλης ουσιαστικής και λειτουργικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορέσει να μας δώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε και αίμα και λεφτά. Η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωση ΝΑΤΟ δεν είναι απλώ επιθυμητή, πιστεύουμε ότι είναι ουσιώδης. Θα ήταν ε, λάθο ε, αν δεν περάσουμε πέρα από τα θα μπορούσαμε και θα έπρεπε τις σχέσεις μας στα μπορούμε και πρέπει. Ε, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τις ε, προκλήσεις της συμπληρωματικότητας, αλλά πιστεύουμε ότι αρκεί Αξίζει τον κόπο να κάνουμε την προσπάθεια. Ένα παράδειγμα. Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα ε, τη στάση του ΝΑΤΟ εξαρτάται από την ικανότητα τη συμμαχία να διενεργεί γρήγορε και αποτελεσματικέ επιχειρήσει ενίσχυση. Η στρατιωτική κινητικότητα είναι βασικό στοιχείο τη άμυνας τη Ευρώπη και πρέπει να εφαρμόσουμε μηχανισμού γρήγορα που στηρίζουν αυτή την ε, προσπάθεια ενίσχυση. Φυσικά χρειαζόμαστε δυνάμει για την ενίσχυση των δυνάμεων που θα είναι εξοπλισμένες, ε, ε, καταρτισμένες και η πρωτοβουλία ετοιμότητας του ΝΑΤΟ ε, θα βελτιώσει πολύ, πολύ έντονα την ετοιμότητα των συμμάχων, των δυνάμεων των συμμάχων. Αυτό είναι θετικό, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μετακινούμε γρήγορα αυτές τις δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη, από την Ευρώπη, προς όλες τις στρατηγικές κατευθύνσεις και να τις συντηρούμε στα θέατρα του πολέμου. Η στρατιωτική κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να ενισχυθεί και τα συμφέροντα και των δύο οργανισμών συγκλίνουν σαφώς εδώ. Τώρα, θα ήθελα να τελειώσω. Η προσπάθεια στεντέρων τη εργασία Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ ε, σε ένα νέο επίπεδο φιλοδοξία είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά με βάση τι κοινέ προτάσει, εάν επενδύσουμε επί τη ουσία και αν δεν ξεχνάμε τις αρχές και τις αρετές του ρεαλισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από τη θεωρία της συνεργασίας πρέπει να περάσουμε στην πραγματικότητα, ειδικά σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή και τακτική συνεργασία. Δέκα λεφτά. Τελειώσανε. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστούμε, στρατηγέ, λέει η πρόεδρος. Ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Γκάλα. Ευχαριστώ για την ε, τοποθέτηση αυτή, την εισήγηση αυτή. Πράγματι, οι 74 δράσεις ε, που έχουμε εντοπίσει είναι η πολλή δουλειά που έχουμε μπροστά μας για να επιτύχουμε συμπληρωματικότητα και προσθέμενη αξία. Η ερώτησή μου είναι ιδιαίτερα επί του τι έχει αλλάξει στην καθημερινή εργασία εντός του ΝΑΤΟ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεδομένης της ε, στάσης του Αμερικανού Προέδρου. Τι κάνετε, περιμένετε τα tweet κάθε πρωί, πώς το χειρίζεστε, δηλαδή πώς έχει αλλάξει η δουλειά. Πόσο δεσμευτικές μπορεί να θεωρείτε τις δεσμεύσεις ε, προς τους Αμερικανούς ή με τους Αμερικανούς και μπορούν να ακυρωθούν επειδή ξύπνησε στραβά το πρωί ο πρόεδρος για να το πω ευγενικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαλέρο είναι ο επόμενος συντονιστής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν σας άκουσα να μιλάτε για την συνθήκη INF και δεν ξέρω αν έχετε και υπόψη σας το ψήφισμα που εγκρίναμε προεβδομάδος θα σας συνέστηνα να το διαβάσετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Θα μας ενδιαφέρει να ακούσουμε ε, τι συζητείτε στο ΝΑΤΟ σχετικά με αυτό το θέμα, τη συνθήκη δηλαδή. Αλλά καθότι προέρχομαι από τη Σουηδία που δεν είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και έχουμε ευρύ πεδίο συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, αλλά όταν είχαμε συνυπογράψει την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων και υποτίθεται ή πετίθεται ότι θα την επικυρώναμε, λάβαμε την απειλή από τον ΝΑΤΟ ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν επικυρώσουμε, θα τερματιζόταν η συνεργασία με τη Σουηδία. Ήθελα λοιπόν από εσά να ακούσω κατά πόσον αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών, των κρατών και αν θεωρείτε ότι πράγματι θα ήταν καλή ιδέα να τερματιστεί η συνεργασία με τη Σουηδία εφόσον δεν επικυρώσουμε. Σας ευχαριστώ. Η Αντιπρόεδρη, ο κύριος Γιάρομιρ Στέτινα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. οι συνάδελφοι, καλύτερα να φορέσετε τα ακουστικά σας για να με ακούσετε θα σας ευχαριστούσα για την ρεαλιστική σας τοποθέτηση και θέλω και εγώ μια ρεαλιστική ερώτηση να σας υποβάλω. Έχουμε την σύγκρουση στην Ουκρανία, πλαίσιο στο οποίο θα έρθετε την εξή ερώτηση. Η ανώτη διοίκηση στην Ευρώπη θα έπρεπε ίσως να εξετάσει το θέμα των συνθήκων της Βουδαπέστης όταν είχε δεσμευθεί η Ουκρανία να αποσύρει τον πυρηνικό της οπλισμό και πολλές και διάφορες χώρες συνεγγυήθηκαν τη συνθήκη εκείνη. Μεταξύ των οποίων και τις Ηνωμένε Πολιτείες δεν θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να ασκήσει μια πίεση σε αυτό ώστε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Και πάλι, σας ευχαριστώ. Η κυρία Μούντι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον στρατηγό για την παρουσία του εδώ και για την παρουσίασή του εδώ. Δύο συνάδελφοι ήδη έθιξαν το θέμα της συνθήκης INF, αλλά θα, πραγματικά θα ήθελα και εγώ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω την απάντησή σας, ιδιαίτερα εν ώψη του, ψηφο, του ψηφίσματος περασμένης εβδομάδος, αλλά και λόγω του αντικτύπου της συνθήκης αυτής στους πολίτες μας, γιατί ήμασταν υπογράφοντες αλλά και βασικοί δικαιούχοι. Κάτι ακόμα που θα ήθελα, που θα με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σας, είναι η θάλασσα του Αζόφ και οι πρόσφατες εξελίξεις εκεί και πώς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Το άλλο ζήτημα είναι αρκετά ευαίσθητο και είμαι σίγουρη ότι θα απαντήσετε και εσείς ευαίσθητα. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν κάποιες πιέσεις, εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ μεταξύ των διαφόρων παικτών και ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε τη δική σας οπτική προκειμένου να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις κοινέ μας θέσεις Και τέλος, και ελπίζω σε ένα πιο θετικό πνεύμα, σχετικά με την, την ε, τη συμπληρωματικότητα εν δράση. Και στο πεδίο το αμυντικό και στο πεδίο το πολιτικό. Θα μπορούσατε να με εξεργαστείτε λίγο περισσότερο το πώς βλέπετε να ενισχύουμε την ενωσιακή συμμετοχή και την όλη δράση αυτήν. Σας ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ στρατηγέ. Ο κύριος Γκάλα ήδη ε, σας ρώτησε για τα tweet του Τραμπ, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι λίγο υπερβαίνει δηλαδή λίγο τα tweet του Πρόεδρου. υπάρχει μια υποψία ότι εν πάση υπάρχει ένας μοχλός εκβιασμού ή πίεσης κατά του Προέδρου. Και στην ουσία αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο που λέμε. Πώς το χειρίζεστε το θέμα αυτό. Μιλήσετε για μια Ρωσία πιο επικίνδυνη. τι σκέπτεστε για την νίκη στην Συρία που τις παραχωρήσαμε όλοι. Ε, την έχει κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη και πιο προκλητική. Και τέλος, ε, και εγώ θέλω να αναφερθώ στις συνέπειες της απόσυρσης των Αμερικανών από τη συνθήκη INF. Τώρα τρομοκρατικές ομάδες στη Συρία και το Ιράκ ε, η ιδεολογία αυτή δεν έχει καθόλου πεθάνει. Έχουμε λοιπόν μια στρατηγική διαλόγου με τους μουσουλμάνους χωρίς τους οποίους δεν γίνεται να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό ο οποίος περνάει από τα αμυντικά συστήματα αλλά και τις κοινωνίες και την συλλογική ψυχολογία. Τι λέτε για το κενό που έχει μείνει επίστηλη Λιβύη. Ο κύριος Ελίμοβιτς λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ στρατηγέ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και το χρόνο που μας αφιερώσατε. Ε, έχω μία ερώτηση για την άποψή σας σχετικά με την παρουσία του ΝΑΤΟ στις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αρκετά τρομακτικά γεγονότα και τάσεις και στην Σερβία και στο Μαυροβούνιο είχαμε και απόπειρα δολοφονίας ενός πρωθυπουργού το οποίο από ό,τι φαίνεται συνδέεται λέει ο μιλητής με τη Ρωσία ή τουλάχιστον με κάποια κέντρα στη Ρωσία Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω για τη δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απόπειρα επιθετική, επιθετικής παρέμβασης στα Δυτικά Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε τον κατάλογο των ερωτημάτων ε, στρατηγέ. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε, να σχολιάσετε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Φοβούμαι ότι ίσω κάποιε από τι απαντήσει μου να είναι απογοητευτικέ. Θα ξεκινήσω με το θέμα του Πρόεδρου Τραμπ. Γιατί το θέσατε κάποιοι. Καταρχά, ω στρατιωτικό διοικητή, ε, αντιλαμβάνεστε ότι οι ερωτήσει αυτέ που θέτει ο Τραμπ είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Και κάποια από την πίεση που διαβιβάζει στο ΝΑΤΟ και στις χώρες μέλη μέσω της προσέγγισής του ε, περνούν και από τους στόχους της αύξησης των αμυντικών δαπανών που έχει θέσει. Νομίζω ότι στην πρόσφατη συνάντηση των Υπουργών Αμήνης ο Αμερικανός Υπουργός ξεκάθαρα εξέφρασε πλήρη στήριξη και δέσμευση προς τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή αν δούμε τις πράξεις και όχι τα λόγια, η αμερικανική υποστήριξη είναι αδιάκοπη. Και χρηματικά και σε επίπεδο αμυντικών εξοπλισμών που έχουν σε ανάπτυξη. Επομένως δεν ανησυχώ καθόλου για την αμερικανική δέσμευση. Υπάρχει μεγάλη απόκληση σχετικά με τα λεγόμενα του Προέδρου, με όποιον τρόπο και τις ε, τελικώς δράσεις της αμερικανικές. Για τις χώρες της Βόρειας Σουηδία και Φιλανδία δεν είχαμε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με Σουηδό εκπρόσωπο. Νομίζω ότι η σχέση είναι εξαιρετική. Και νομίζω ότι το σχέδιο δράσης να αναπτύξουμε μια καλύτερη προσέγγιση ο ένας του άλλου και κατανόηση αμοιβαία είναι θετική. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία, κανένας συσχετισμός μεταξύ αυτού του επίπεδου και της οποιασδήποτε επικύρωσης της INF. Και εκπλήσωμε από αυτό που λέτε γιατί δεν το έχω δει στη δουλειά που κάνω εγώ προσωπικά. Εγώ θα έλεγα ότι τα πράγματα πάνε καλά. Για τη συνθήκη της Βουδαπέστης του 1984 για την Ουκρανία είναι πολιτικό ζήτημα. Η Ουκρανία βεβαίω δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Υπάρχει η δέσμη στήριξης προς τη χώρα αυτή, αλλά θα παραμείνει το ζήτημα αυτό δύσκολο και περιπλοκό και σε επίπεδο συμμαχία και σε επίπεδο υλοποίηση και θα τοποθετούσα και τη θάλασσα του Αζόφ στο ίδιο αυτό πεδίο. Ε, το ΝΑΤΟ είναι μια συνενετική συνεργασία των 29 και η θάλασσα του Αζόφ οπωσδήποτε είναι σε πολιτικό και όχι στρατικό αμυντικό επίπεδο. Τώρα εγώ αυτό που έχω δει στο ΝΑΤΟ είναι ότι έχουμε περάσει και στο παρελθόν δυσκολίες και παρά τα σκαμπανεβάσματα της πολιτικής στην Ευρωακή Ήπειρο, οι σχέσεις, οι αμυντικές, οι σχέσεις των μελών είναι καλύτερες. Και σε γενικές γραμμές υπάρχει κατανομή άχθους και ευθύνης και σε όλα τα σημεία κρίσης όλα τα μέλη προσπαθούν να κοιτούν τα πράγματα και από την οπτική των άλλων μελών. Αν δείτε την πρόοδο που έχουμε ε, σημειώσει από το 2014 μέχρι τώρα με το σχέδιο τιμότητας, με την αυξημένη θαλάσσια παρουσία, με τους νέους δίκτες, ε, τα προγράμματα αποτροπής ε, και τις πρωτοβουλίες ετοιμότητας, αυτή η συμμαχία δεν μοιάζει καθόλου διαρρεμένη θα έλεγα εγώ μοιάζει πολύ ενωμένη στα δικά μου τα μάτια. Για τις τρομοκρατικές ομάδες συμφωνώ ότι ε, βασιζόμαστε ευρέως σε χώρες ε, συνεργάτες Βεβαίως δουλεύουμε στα πλαίσια της ε, οικοδόμηση σταθερότητα, αλλά πρόκειται για μια περιοχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πράγματι θα μπορούσαν μάλλον να κάνουν περισσότερα. Για τη συνθήκη INF, και είδατε και τη δήλωση των Υπουργών Αμήνη. σχετικά με την Αμερικανική γραμμή για την συνθήκη, αν δεν την έχετε δει μπορώ να σας την ε, διαβιβάσω, αλλά δεν θα είχα κάποιο άλλο σχόλιο να κάνετε. Για τη Συρία Συμφωνώ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και βεβαίως είναι μια επιχείρηση συμμαχίας και όχι του ΝΑΤΟ, παρότι κάποιες χώρες μέλη συμμετέχουν και για τα Δυτικά Βαλκάνια τέλος. Αυτή τη στιγμή, όπως θα ξέρετε, είμαι διοικητής της ε, επιχειρησιακής μονάδας για τη Βοσνία για τους ε, τους 6.000 που υποστηρίζουν τα, τις επιχειρήσεις K4 στο θέατρο αυτό επιχειρήσεων και σε γενικές γραμμές υπάρχει συμφωνία και ανησυχία για την κατάσταση της ασφαλείας Ανατολικών Βαλκανίων. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ στενή συνεργασία και προσπάθεια να συνοδεύσουμε τις χώρες αυτές σε μια πιο σταθερή κατάσταση, αλλά γνωρίζετε και εσείς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην ε, Βοσνία και όπως είπε και είπατε εκπρόσωπος ε, ε, υπάρχει αυτή η μαζική φυγή νέων ανθρώπων από τη Βοσνία πρέπει να κάνουμε περισσότερα και στο ΝΑΤΟ πραγματικά διερευνούμε το πώς μπορούμε με μεγαλύτερη συνέπεια να δρούμε, αλλά βραχυπρόθεσμα δεν ξέρω αν όλα αυτά θα επιφέρουν κάποια εντυπωσιακή αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε σημαντικές ερωτήσεις μετά τις απαντήσεις αυτές, διευκρινιστικές προς τον στρατηγό. Έχουμε χρόνο για λίγες ερωτήσεις ακόμα. Κύριος Γκάλερ, μια γρήγορη. Αναφερθήκατε στην αποστολή Αλθέα, που είναι η τελευταία κοινή αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ στη Βοσνία. Και το συζητήσαμε και με κάποιον άλλο μιλητή το πρωί. Υπάρχουν κάποιες ανατρεπτικές δυνάμεις και κάποιες ταραξίες στην Βοσνία που θέλουν να τερματίσουν το status quo. Και ρωτώ, επειδή εκεί είμαστε πολύ περιορισμένοι, στη Βοσνία, αλλά έχουμε σε επιφυλακή κάποιους εκτός Βοσνίας, κοντά. Αυτοί εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενισχύσουν τις δυνάμεις αυτές στη Βοσνία, σε περίπτωση που ο συνήθις ύποπτος θέλει να ε, οδηγήσει σε ταραχές και να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε. Για να απαντήσω σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να κατανοεί ο κόσμος ε, ότι έχουμε μόνο 610 παντού. Είναι πολύ μικρό αυτό το αποτύπωμα, το ε, ε, ε, ίχνος που αφήνουμε. Αλλά κάνουμε ασκήσεις κάθε χρόνο για τις ενισχύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν. Και πρόσφατα είχαμε για ένα τρίμηνο κατά τη διάρκεια των εκλογών παρουσία. Ξέρουμε και έχουμε μηχανισμό ελέγχου εκεί και με το Βερολίνο ΣΥΝ. Εγώ συντονίζω τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ και θα μπορούσαν από την ΚΕΙΦΟΡ να αποσπαστούν κάποιες δυνάμεις για να υποστηρίξουν ε, τη δύναμη στη ε, Βοσνία. Η κυρία Κλέρ Μούντι. Ευχαριστώ πολύ. Αφού μας δώσατε περισσότερο χρόνο για ερωτήσεις, αμέσως μου ήρθαν ερωτήσεις. Μοιραία και αναπόφευκτα. Ε, ένα πιο συγκεκριμένο θεματικό. Τι γίνεται με τις γυναίκες στην ασφάλεια και την ειρήνη. Ξέρω ότι το ΝΑΤΟ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σχετικά. Εσείς πώς το βλέπετε. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σας για την δυνατότητα του ΝΑΤΟ και την ικανότητα του ΝΑΤΟ να έχει μια στρατηγική με βάση το φύλλο. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Ε, λοιπόν, όταν ανέλαβα, ε, ήμουν ε, πρωταθλητής ε, επί μία πενταετία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2016 για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Υπάρχει και σύμβουλος διορισμένος στην ομάδα διοίκησης για θέματα ισότητας και φύλου και γνωρίζω ότι και το ΝΑΤΟ προσπαθεί να υλοποιήσει τον ίδιο στόχο. Και εγώ ως αρμόδιος ε, στο ΝΑΤΟ προσπαθώ να το βάλω και ως προϋπόθεση και ως κριτήριο να υπάρχουν σύμβουλοι για το φύλλο. Ε, πάντως δεν ισχύει αυτό σε όλες τις χώρες, δεν υπάρχει. Και χρειάζεται φυσικά πάρα πολύ ε, μεγάλη εκπαίδευση. Καλό είναι να έρχονται εκπαιδευμένοι και έτοιμοι ε, βλέπω βελτιώσεις τους επόμενους μήνες, αλλά και πάλι αυτό με συναρπάζει. Ε, μια συμμαχία 29 κρατών και βλέπουμε ότι οι χώρες διαφέρουν ως προς το επίπεδο ισότητας των φύλων. Δεν είναι καθόλου ίση αυτή η κατάσταση. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο για να σας βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Η πρόεδρος, για να διευκρινίσω κάτι, η Κλέρ Μούντι είναι αρμόδια στο διευρυμένο Προεδρείο μας ε, που ασχολείται με αυτά τα θέματα και με αυτά τα. Η απάντηση είναι καταφατική, διότι τα κράτη είναι εκείνα που απαρτίζουν τον ΝΑΤΟ και κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς αποφασίζετε ε, τι θα ζητήσετε από εμά. Και αν έρθει ένα πολιτικό μήνυμα στεναρό ότι θα πρέπει σε επίπεδο διοίκησης παντού όλες οι μονάδες να έχουν ένα σύμβουλο για θέματα φύλου, θα υλοποιηθεί. Αλλά αυτό εξαρτάται από τη χώρα. Ε, κάποιες χώρες είναι πολύ προηγμένες σε θέματα ε, διαφορετικότητας ε, και φύλου. Ορισμένες τώρα μόλις να καλύπτουν αυτό το έδαφος. Οι στρατιώτες διαταγές υπακούν. Αν έρθει η διαταγή, εμείς θα την εκτελέσουμε. Η Πρόεδρος, έχω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση και μάλλον θα είναι και η τελευταία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Πώς το αξιολογείτε αυτό, τα επιτεύγματα στο συγκεκριμένο κλάδο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο χώρος αυτός ο κυβερνοχώρος και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην άμυνα, την κυβερνοάμυνα. Ξέρω ότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που συνεργάζονται με ρωτάνε για την επίθεση, τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, όχι στην άμυνα. Η επίθεση είναι πιο περίπλοκο. Το εντάσσουμε και αυτό στα σχέδιά μας, εκτός από την άμυνα, αλλά ποτέ δεν έχω δει ευρωπαϊκή αποστολή που να έχει ζητήσει τέτοια δυνατότητα, να έχουμε τη δυνατότητα επίθεση στον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ. Όπως πάντα, συναρπαστική ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας βλέπουμε πιο συχνά στο προσεχές μέλλον. Και μπορείτε να υπολογίζετε στην ε, σύσφυξη των δεσμών και με το SHAPE. Παρακαλώ να χειροκροτήσουμε τον στρατηγό. Thank Θα αρχίσουμε με το επόμενο σημείο. Πάρα αυτά, παιδιά. Good afternoon. Grüßen Sie. Schön, dass Sie gekommen sind. Nee, nee, bin ich nicht. Ich bin sein Kollege, der Herr Schröder. Ich bin sozusagen hier für das Sekretariat. So the others okay. will arrive. We still have about seven minutes to go. How do you pronounce this name I ask you yeah. about? I will find this out now. I, will find this out. I think it's a Frenchman of, let's say, slightly oriental. Yeah. So probably.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

Ladies and gentlemen, please be seated. Καθίστε παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Τελευταίο σημείο της σημερινής μας συνεδρίασης. Τελευταίο ουσιαστικό σημείο είναι η κοινή δύναμη των πέντε χωρών για τη Σαχέλ στο Μαλί. Θα μιλήσουμε για την ασφάλεια και τα ανθρωπιστικά θέματα στο Σαχέλ. Και τι κάνουν οι, χώρες, οι πέντε χώρες Σαχέλ. Είναι πολύ επίκαιρο θέμα. Πρέπει να αποφασίσουμε για τη μελλοντική εντολή που θα εκπνεύσει σύντομα. Υπάρχουν ε, εξελίξεις στην ασφάλεια. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τους ομιλητές μας. Τέσσερα άτομα. Θα σας τους παρουσιάσω σε λίγο. Μάλλον θα πάρουν το λόγο σε λίγο. Τώρα θα τους παρουσιάσω. Αριστερά μου είναι ο πρώτος ομιλητής, ο κύριος Ιρσάντ Ραζάλη, τμήματάρχης για τη Δυτική Αφρική στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Μαρκ Σταλμάντς, επικεφαλής του τομέα για τις χώρες Σαχέλ στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αμέσως ε, δίπλα η κυρία Σιμών Σνάμπελ, ερευνήτρια, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο της Φραγκφούρτης για την Ειρήνη. Μετά, κατά τις παρουσιάσεις, μπορεί να έρθει και ο κύριος Ρόρι Κίν. Αλλά δεν είναι σίγουρο. Γι' αυτό δεν την υπολογίζω αυτή την παρουσίαση και χωρίς πολλά πολλά θα δώσω το λόγο στους διακεκριμένους ομιλητές με την ίδια σειρά στον κύριο Ισάντ Ραζάλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Καλημέρα. Θα σας παρουσιάσω κάποια πράγματα. Τρία λεπτά έχουμε μόνο, να το πω αυτό στην αρχή. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία... να θέσω το πολιτικό πλαίσιο για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις πέντε χώρες Σαχέλ γενικά και της ευρωπαϊκής στήριξης ε, στην, στο να μπορέσει να γίνει επιχειρησιακή η κοινή δύναμη των χρόνων Σαχέλ. Η Σαχέλ έχει μια κρίση παλιά θα έλεγα. Η κατάσταση το 2012-2013 επιδεινώθηκε όταν το Μαλί ε, δέχτηκε επίθεση από τρομοκράτες και εξτρεμιστές και αυτό προκάλεσε αντιδράσεις στρατιωτικές από τους Γάλλους και δημιουργήθηκε ή μετασχηματίστηκε η Μίσκα ε, από επιχείρηση για την Αφρική σε επιχείρηση του ΟΗΕ ε, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της ε, χώρας αλλά και για να εγγυηθεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες που ε, υπογράφτηκαν μεταξύ κάποιων δυνάμεων του Μαλή, της κυβέρνησης και εκπροσώπων των ενάπλων δυνάμεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρέμβασή μου λοιπόν και το 2015 οι πέντε βασικές χώρες ε, της περιοχής ε, του Σαχέλ, το Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, ο Νίγηρας, με το Τσάντ και τη Μαυριτανία, πήραν την πρωτοβουλία και είπαν ότι πολιτικά είχαν κάθε συμφέρον να πολεμήσουν μαζί ένα κοινό εχθρό που ήταν οι τρομοκράτες, οι τρομοκρατικές απειλές. Αυτή η δραστηριότητα περνούσε μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας μιας κοινή δύναμης, δηλαδή μιας στρατιωτικής δύναμης που θα δημιουργούσαν αυτές οι πέντε χώρες του Σαχέλ και που θα αποτελείται από τάγματα τα οποία θα ήταν στη διάθεση της περιοχής ε, και θα την αποτελούσαν ε, τμήματα δυνάμεις των πέντε χωρών. Προστιθέμενη αξία υπήρχε σε σχέση με τις ε, εθνικές ενόπλες δυνάμεις που πολεμούσαν μόνες τους, ε, περιπολούσαν στα συνοριακά, συνοριακές περιοχές και είχαν δικαίωμα να δώσουν συνέχεια όταν δίωκαν ε, τρομοκράτες. Είτε από τη μία είτε από την άλλη μεριά των συνόρων. Μπορούσαν δηλαδή να δραστηριοποιηθούν και προ τι δύο μεριέ των συνόρων. Αυτή ήταν η προσθέμενη αξία. Από το καλοκαίρι του 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είπε ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία που όπως σας είπα είχε το βασικό πλεονέκτημα ότι ήταν καρπός πολιτικής βούλησης αυτών των πέντε χωρών και θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μια σημαντική ένδειξη δέσμευσης καταρχά των πέντε χωρών και δεύτερον σε επιχειρησιακό επίπεδο οι προσπάθειες και οι δυνάμεις ε, που κινητοποίησαν η διεθνής κοινότητα και οι χώρες αυτές ε, δεν ήταν σε θέση να μειώσουν τρομοκρατική απειλή. Ακριβώς γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είπε ότι θέλει να υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία. Τον Ιούλιο του 2017 η κυρία Μογκερίνη επιβεβαίωσε αυτή την υποστήριξη σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο κινητοποίησε 50 εκατομμύρια ευρώ για να εξοπλίσει την κοινή αυτή δύναμη τον Φεβρουάριο του 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση οργάνωσε μια διάσκεψη για την υποστήριξη ε, των πέντε χωρών της ΑΧΕΛ, κυρίως υπέρ της κοινή αυτής δύναμης, που είχε πει ότι χρειάζεται 300 εκατομμύρια ευρώ περίπου για τις ανάγκες της. Ε, η διάσκεψη αυτή ακριβώς έγινε για να εξασφαλιστεί αυτό το ποσό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσέφερε 50 επιπλέον εκατομμύρια ε, σε εκείνη τη διάσκεψη για να εξασφαλιστούν τότε και να ικανοποιηθούν κάποιες ανάγκες, κυρίως ε, σε επίπεδο εξοπλισμού. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι αυτή η διάσκεψη όμως έγινε λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες μετά την υιοθέτηση ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ το 23 κάθετος 411 που πρόβλεπε μεταξύ άλλων την ε, κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, όπως είπα, την εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός ε, μηχανισμού συντονισμού των αναγκών και των προσφορών ε, για την κοινή δύναμη και την υποστήριξη στην ανάπτυξη στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιχειρήσεων από αυτή την κοινή δύναμη. Ένα από τα βασικά μελήματα που υπήρχαν τότε ήταν ότι θέλουμε συλλογικά να στις ζώνες που δεν καλύπτουν, ας πούμε, που δεν καλύπτει το, οι κρατικές δυνάμεις του, του, του Μαλή, να επαναδιατρανώσει το κράτος την παρουσία του. Επίσης, η κοινή δύναμη, χάρη στις επιχειρήσεις της, να σταματήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό ακριβώς σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ΟΗΕ, μαζί με την έγκριση ε, των κρατών, των πέντε κρατών δηλαδή της ΑΧΕΛ και με, τις, ε, την έγκριση των κρατών της Αφρικανικής Ένωσης, ε, συμφωνήθηκε να υπάρχει αυτό το πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το σεβασμό του διεθνούς ε, δικαίου. Υιοθετήθηκε λοιπόν και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται από την κοινή δύναμη G5. Με τη βοήθεια ε, του ΟΗΕ και του Γραφείου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτά προς το παρόν. Σταματώ εδώ εγώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Στάλμανς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ στα γαλλικά θα μιλήσω. Για να συμπληρώσω, λοιπόν, ε, τα όσα είπε ο συνάδελφος από την ΙΕΔ, Ήθελα να πω ότι η δράση της ε, Κομισιόν ε, στο πλαίσιο των πέντε χωρών είναι στρατιωτική, μεν, αλλά ακολουθεί την κατεύθυνση και της ανάπτυξης εκτός της ασφάλειας. Επομένως, σε όλη αυτή την ευαίσθητη ζώνη, στην Μπουρκιναφάσο, σε κάποιες περιοχές του Νίγηρα και του Τσάντ, δεν μπορούμε πλέον να καταβάλουμε προσπάθειες ανάπτυξης όπως τις κάναμε στο παρελθόν, διότι έχει περιπλακεί η κατάσταση ασφαλείας και δυσκολευόμαστε να βρούμε φορεί που να μπορούν να λειτουργήσουν, να εργαστούν στην περιοχή αυτή, λόγω της απειλής που υπάρχει. Επομένως, ανάπτυξη αλλά καλά πλαισιωμένη σε επίπεδο ασφαλείας, με πολύ προσοχή στις τοπικές ε, κοινωνίες γιατί δεν αποστέλνουμε μόνο στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια και άλλη βοήθεια. Γιατί στο σύνολο της ενίσχυσης μιλούμε για 4 δισεκατομμύρια για τις πέντε χώρες για την περίοδο 2014-2020. Από τα 4 αυτά δισεκατομμύρια το τμήμα ασφάλειας, το στρατιωτικό, η στρατιωτική δαπάνη ήταν το 2 με 5% τα υπόλοιπα ήταν αναπτυξιακά κονδύλια και ανθρωπιστικής βοήθειας. Επομένως είναι σημαντική, σημαντικός αυτός ο συσχετισμός. Είναι σημαντικός για εμάς και υπό τη γεωπολιτική έννοια, δεδομένη της σημασία του G5 των πέντε χωρών, προκειμένου όλα μας τα μέσα που έχουμε διάθεσή μας να μπορούν να ενεργοποιούνται για να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις περιοχής. Μιλούμε για χρηματοδότηση για την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανεξιακή βοήθεια, την εσωτερική ασφάλεια και τη χρηματοδότησή της, την αμυντική ενίσχυση, την επιστροφή των τοπικών αρχών και τις μεταναστευτικές ροές, όλα αυτά στην ίδια γεωγραφική ζώνη. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί, ενεργοποιώντας όλα μας τα μέσα, όλα μας τα κονδύλια για να αντιμετωπίζουμε διαρθρωμένα τις ανάγκες και τις προκλήσεις. Για να συνεχίσω τώρα την ε, αναφορά στην ε, κοινή αυτή ε, ομάδα τη στρατιωτική της περιοχής καλείται να αντιμετωπίσει τα θέματα αμήνης με σώματα στρατιωτικά και από τις πέντε χώρες γιατί οι επιχειρήσεις Μπάρκαν και μίνουκμαν ε, κατευθύνονται από άλλες χώρες. Είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν δράσεις και οι ίδιες οι πέντε χώρες. Είχαμε μια ενίσχυση 5 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι εδώ. Εξετάζουμε και την αύξησή της λόγω της επιδείνωσης κατάστασης ε, ασφάλειας ή στην ε, Μπουρκίνα Φάσο. Μιλούμε κυρίως για εξοπλισμό ενίσχυση της μόνιμης ε, γραμματείας ε, του G5, τα θέματα συμβατότητας ε, των συστημάτων και η συμμόρφωση με τα προς τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το κύριο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής και για τις πέντε χώρες που έχουν επικυρώσει το πλαίσιο αυτό για τις θερατικέ δυνάμεις εκτός της Μπουρκιναφάσου αλλά πιέζουμε τη χώρα αυτή να επικυρώσει και για τις δικές της στρατιωτικές δυνάμεις. Για τον εξοπλισμό τον ίδιο. Ίσως να υποτιμήσαμε λίγο τον χρόνο που θα χρειαζόταν η θέση σε ετοιμότητα αυτής της ε, κοινή δυνάμεως και για μας και για την, ε, στην Devco είναι ένα ε, νέο αντικείμενο αυτού του είδους η πρωτοβουλία στον χώρο τον αμυντικό Υποτιμήσαμε λοιπόν το χρόνο που χρειαζόταν για να υπάρξει ένας εξορθολογισμός, όπως και ο απαραίτητος χρόνος για την παράδοση του στρατιωτικού εξοπλισμού. Ήμασταν ίσως λίγο υπερβολικά αισιόδοξοι, όπως ήμασταν ε, κάπως αισιόδοξοι και για την ικανότητα των χωρών αυτών να συμφωνούν, να έχουν μια κοινή δομή στρατιωτικής διοίκησης υπερτιμήσαμε επίσης ε, τις ικανότητες, τις δυνατότητες της μόνιμης γραμματείας του G5 για την γραμματιακή υποστήριξη αυτής της κοινής δυνάμεως. Αυτό δεν θα μας αποτρέψει από το να επιτύχουμε τους βραχυπρόθεσμους στόχους μας. Ε, θα μείνω εδώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Σίμων Σνάμπελ, που είναι ερευνήτρια στη Φραγκφούρτη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση στην υποεπιτροπή σας. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ για να σας ε, ε, παρουσιάσω τις απόψεις μου και τις σκέψεις μου για την συνεργασία ε, G5 στο Σαχέλ, γιατί εργάζομαι ε, για αυτό το τομέα και κάνω έρευνα εδώ και χρόνια. Θα επικεντρωθώ σε δύο στοιχεία. Πρώτον, ε, στις τρέχουσες προκλήσεις ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη συνέχεια θα θέσω αυτή την πρωτοβουλία των πέντε του Σαχέλ στην ε, Άψα που είναι η Αφρικανική Αρχιτεκτονική για την Ειρήνη και την Ασφάλεια για τη διαχείριση των κρίσεων και των συγκρούσεων. Ε, δημιουργήθηκε αυτή η δύναμη των πέντε χωρών ε, για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία, να ενισχύσει τη φύλαξη των συνόρων, να προλαμβάνει τα λαθρεμπόρια και να επαναφέρει την κρατική αρχή. Είναι προβληματική αυτή η προσέγγιση, γιατί δεν ξέρουμε ε, ποιοι είναι οι στόχοι. Δεν είναι ένας ο εχθρός, είναι δεκάδες οι ένοπλες δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές οι τρομοκρατικές δυνάμεις και ε, η πρώτη ενέργεια ε, πρέπει να είναι η ταυτοποίησή τους και ο διαχωρισμός από τον άμεχο πληθυσμό. Μήπως να μην διαβάζετε τόσο γρήγορα, λέει η Πρόεδρος, για να σας μεταφράζουν. Δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Έλεγα λοιπόν ότι είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι στόχοι και να διαχωριστούν από τον άμαχο πληθυσμό ε, και είχε και συνέπειες απροσδόκητες. Όπως γνωρίζουμε, ε, ε, ένοπλες δυνάμεις του μαλί και της Μπουρκίνα Φάσο εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκτελέσεις, εξαφανίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις. Διαβάζετε πάρα πολύ γρήγορα Ε, γενικότερα οι ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή ε, γενικά παραδοσιακά επιτίθενται σε άμαχους, ιδιαίτερα στο κεντρικό και βόρειο Μαλί και αυτό υποδαβλίζει τις ε, τοπικές συγκρούσεις μεταξύ γεωργών και νομάδων. Αλλά γενικώ ακόμα και όταν δεν είναι βίαιοι, δεν έχουν υποστήριξη από τις ένοπλες δυνάμεις τους, από τις χώρες τους και γενικά εμφανίζουν ε, κρούσματα διαφθοράς και εγκληματικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Άρα λοιπόν ε, θα ε, συστήσω στο τέλος της παρέμβασής μου να συσταθεί επιγόντως και μια πολιτική μονάδα που θα συνοδεύσει τη στρατιωτική. Έρχομαι στο δεύτερο στοιχείο δεν λειτουργούν στο κενό αυτές οι ενοπλές δυνάμεις, αλλά ε, σε ένα σύνολο περίπλοκων ε, θεσμών και θεσμικών οργάνων. Και κινδυνεύουν τώρα να δημιουργήσουν μια παράλληλη δομή, παράλληλη προς την ε, αρχιτεκτονική ασφαλείας άψα. Μέχρι στιγμής τι βλέπουμε. Η Αφρικανική Ένωση καταβάλει προσπάθειες ε, να αναπτύξει μια κοινή στρατιωτική δύναμη. Είναι η ASF, μια δύναμη σε επιφυλακή, ένα είδος εφεδρείας που συνιστούν τα κράτη-μέλη ε, και είναι έτοιμη να επέμβει ε, όταν χρειάζεται. Υπάρχουν πέντε περιφέρειες, η Βόρεια Αφρική, η Δυτική, η Κεντρική, η Ανατολική και η Νότια και θα πρέπει να έχει μια επιχειρησιακή τέτοια μονάδα επιφυλακή το 15, ήδη από το 15 ουσιαστικά, μόνο στη Δυτική Αφρική έχει γίνει αυτό και έχουν αναπτυχθεί στην παρέμβαση μετά τις εκλογές στην Κάμπια και πρόσφατα στο Μάλι ε, και παλαιότερα το 2012. Ωστόσο, η εμπειρία στο Μαλί έδειξε ότι ε, δεν ανταποκρίνεται αυτή η οργάνωση στις ε, περιφερειακές και τοπικές προκλήσεις που γνωρίζει το Ομαλή γιατί είναι κάποιες ε, περιφερειακές ταξιαρχίες προκαθορισμένες. Επειδή λοιπόν δεν εφαρμόζεται σωστά αυτό το σύστημα, ε, δεν μπορεί η χώρα και η γενικότερα περιοχή να ε, ανταποκριθεί. Γι' αυτό δημιούργησαν την αφρικανική δυνατότητα για άμεση απόκριση, ΑΣΕΡΚ. έδειξε η εμπειρία ότι δεν πρόκειται ποτέ αυτή η μονάδα να λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί. Ε, άρα η ομάδα των πέντε κρατών ε, είναι άλλη μία στρατιωτική δύναμη στην Ήπειρο και το Αρμόδιο Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης ε, αποφάσισε να ενταχθεί ε, παράλληλα με άλλες δομές όπως είναι η MNJTF, η πολυεθνική δύναμη ε, και άλλα στοιχεία της αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει η προσπάθεια αυτή. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη διαδικασία θεσμοθέτησης και επίσημης συγκρότησης. Ωστόσο, ε, η MNJTF σε αντιδιαστολή με το G5. Είναι κάτι διαφορετικό. Το MNJTF ασχολείται με τις περιοχές που έχει παρουσία η οργάνωση Boko Haram. Η Αφρικανική Ένωση ε, δίνει στρατιωτική, μάλλον ε, επιμελητεία και υποστήριξη εφοδιαστική, ε, ενώ η χρηματοδότηση είναι από τα κράτη-μέλη αυτό έρχεται να περιπλέξει και να κατακαιρματίσει ακόμα περισσότερο την αρχιτεκτονική. Γι' αυτό σας προτείνω τις εξής συστάσεις σε ό,τι αφορά ε, την ε, πολιτική διαδικασία εσωτερική και εξωτερική θα πρέπει να υποστηριχθεί κοινή δυναμία, αλλά υπάρχει κίνδυνος να έχουμε παράλληλε δομές, διαδικασίε και ικανότητε, αντί να έχουμε εναρμόνιση και συνέργειες για τη διαχείριση των κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει στρατηγική συμβουλή για να εναρμονιστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης και οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες εντός της αρχιτεκτονικής άψα. Επίσης, χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο ε, σε όλη την Ήπειρο και έχει ρόλο η, Ευρω... η Αφρικανική Ένωση να διαδραματίσει εκεί για την ομάδα των πέντε. Ε, είπα και στην αρχή ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ε, ένα πολιτικό σκέλος να έρθει να συμπληρώσει το στρατιωτικό στην ομάδα G5 θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο τόπιος πληθυσμός στην προσέγγιση αυτή και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για να υπάρχει εμπιστοσύνη και για να εμπλέκεται ο πληθυσμό. Η Μινούσμα και οι αποστολές εκπαίδευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να ε, έχουν και αυτές μια πολιτική διάσταση για να μοιράζονται εμπειρίε, να ανταλλάσσουν πληροφορίες κτλ. Ας πούμε σχολεία ε, ε, ειρηνευτικά. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τα ε, κράτη ε, G5 στο Σαχέλ θέλουν να δημιουργήσουν δικά τους κέντρα εκπαίδευσης. Επίσης, θα πρέπει να ακούσουν και τι λέει η Αφρικανική ε, Ένωση και οι παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γενικά τους δέχεται ο πληθυσμός και θεωρεί ότι χρειάζονται αλλά κάποιο πρέπει να τους παρακολουθεί, ιδιαίτερα εκεί που δεν φτάνουν οι παρατηρητέ των Ηνωμένων Εθνών. Χρειάζεται υποστήριξη του αμάχου πληθυσμού για να αυξηθεί και η αξιοπιστία και η ε, συνεργασία εκεί ε, της μονάδας αυτής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να σας συστήσω κάποιον που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί είχαμε την ευκαιρία να τον υποδεχθούμε στην αρχή της θητείας είναι ο κύριος Κίν ο οποίος είναι επικεφαλής ε, του Γραφείου Συνδέσμου των Ηνωμένων Εθνών ε, στις Βρυξέλλες και ασχολείται με θέματα ειρήνης και ασφάλειας. Θα θέλαμε να επωφεληθούμε από την ευρύτατη γνώση της περιοχής που έχει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Κίν. Σας ευχαριστώ αξιότιμη κυρία Πρόεδρε Φωτίγκα. Με χαρά επιστρέφω στην υποεπιτροπή σας. Και με χαρά βρίσκομαι εδώ με τα αξιότιμα μέλη, το προσωπικό, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα άλλα μέλη του πάνελ σας. Σας ευχαριστώ που τοποθετήσετε το θέμα αυτό στην Μυρίσια διάταξη γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε μιλήσει αρκετά για θέματα πολυμέρειας και για την ανάγκη ε, ευρεία συνεργασίας αλλά και στενή συνεργασίας Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωση. ανάγκη που είναι μια πραγματικότητα ιδιαίτερα κοιτώντα την περιοχή του Σαχέλ. Το την κοινή αυτή δύναμη των πέντε χωρών μέσω του σχεδίου προτεραιότητος, μέσω της συμμαχίας για το Σαχέλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη συνεργάζονται πολύ στενά προς την κατεύθυνση αυτή, μαζί με τον συνάδελφο στα αριστερά μου, αλλά και του συναδέλφου στη Νέα Υόρκη, σε πολλές από τις πτυχές του πράγματος αυτού και ήθελα να τονίσω από την αρχή ότι το πιο σημαντικό είναι οι πρακτικές λεπτομέρειες. Γιατί οι ρητορικέ τοποθετήσει είναι εύκολε, αλλά στην πρακτική συνεργασία αντιλαμβάνεται κανείς πόσο καλά πρέπει να συνεργαστεί στην περιοχή του Σαχέλ, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά και περίπλοκα. Χρειάζεται λοιπόν αναπτυξιακή βοήθεια και βοήθεια σε επίπεδο διπλωματίας προς τις χώρες αυτές. Η άλλη πτυχή που είναι ενδιαφέρουσα να σημειώσει κανείς ε, εδώ είναι το επίπεδο της δέσμευσης, της συμμετοχής. Μιλούμε για τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζουν μια περιφερειακή πρωτοβουλία. Αλλά η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι των Ηνωμένων Εθνών και δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι Τη γεωγραφική αυτή της και εμείς κοιτούμε πώς καλύτερα μπορούμε να βοηθήσουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το υπογραμμίσει κανείς. Τώρα, για τις πρακτικές πτυχέ, στι οποίε ήδη αναφέρθηκα, για την κοινή δύναμη G5 και το που βρισκόμαστε. Ε, πρόκειται για μια έντολη περίπλοκη που θα έχει και καθήκοντα δύσκολα. Εμείς θα παραμείνουμε εστιασμένοι και θα υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή σε όλη της την τροχιά. Δεν μπορούμε να ξεχαστούμε, πρέπει να συνεχίσουμε την παρακολούθησή μας και την υποστήριξή μας. Και γι' αυτό συναντήσεις όπως σημερινή είναι πολύ σημαντικές. Την Προεδρία του G5 έχει αυτή τη στιγμή η Μπουρκίνα Φάσο, χώρα η οποία ε, επιθυμεί ιδιαίτερα να οικοδομήσει και τη μόνιμη γραμματεία στην Νουακτσότ, μια γραμματεία που να είναι τελικώς λειτουργική και αποτελεσματική. Υπό την έννοια αυτή τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποστηρίξει τον ε, τακτικό γραμματέα του G5 και μέσω της παρουσίας μας ε, του Γραφείου Συνδέσμου για τη Δυτική Αφρική και το Σαχέλ που βρίσκεται στο Ντακάρ έχουμε εγκαταστήσει και μία παρουσία συνδέσμου στην Νουακτσότ για να συνεργαστούμε με την μόνιμη αυτή δομή, την γραμματεία και ανά τρεις μήνες έχουμε μετακύληση προσωπικού και από το Μαλή ώστε να υποστηρίξει το προσωπικό αυτής της δομής του G5. Και στην Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε την συνεχιζόμενη δέσμευσή της και την υποστήριξή της και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί. Τώρα, στο συγγνώμη αν ε, αναφέρθηκε ήδη και ζητώ συγγνώμη καθυστέρησα γιατί χάθηκα λίγο στους διαδρόμους, ότι υπήρχε ε, μία κοιλιά στην εντατικότητα της ε, δραστηριότητας αυτής και αυτό οφείλεται στην επίθεση που έγινε στην έδρα, ε, στο αρχηγείο της κοινή δύναμης και έπρεπε να πάμε από την Σαβέρε στην Μπαμάκο Όλα αυτά χρειαζόταν και χρόνο, υπήρχε και εκλογική διαδικασία στο Μαλί. Ε, όλα αυτά οδήγησαν σε άλλα συνδεδεμένα προβλήματα, αλλά η κοινή αυτή δύναμη επανήλθε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ιδιαίτερα στο τρίγωμο Πιτάκου Γκούρμα, αν ακούσαμε καλά τον ομιλητή, τον Ιανουάριο, και για να επανέλθω και στο πνεύμα της πολυμέρειας που ανάφερα στην αρχή, η Μινούσμα υποστηρίζει την κοινή αυτή δύναμη G5 υπό το ψήφισμα 2391 των ΕΕ. Ψήφισμα στο πλαίσιο του οποίου η Μινούσμα έχει παράσχει βοήθεια, εξοπλισμό και οργανωτική ενίσχυση ή ε, ε, στην αποστολή. Και στο πλαίσιο των πρόσφατων αυτών επιχειρήσεων που σας ανέφερα τον Ιανουάριο. Η Μινούσιμα βεβαίως αναγκάστηκε να απορρίψει αιτήματα τροφίμων και καυσίμου για την δύναμη που επιχειρούσε εκτός του Μαλή, γιατί υπό το ψήφισμα 2391 η Μινούσμα μπορεί να παράσχει τεχνική αρρωγή και υποστήριξη, και το οποίο το περιγράφει και το περιορίζει αυστηρά το ψήφισμα για επιχειρήσεις εντός του Μαλή. Η Μινούσμα όμως δεν έχει εντολή για υποστήριξη ε, ε, επιχειρήσεων εκτός των συνόρων της χώρας. Εξού και είναι σημαντική η πολυμέρεια. Άλλη μια ενδιαφέρουσα πτυχή του ψηφίσματος 2391 είναι ότι έθεσε έναν ιδιαίτερα καινοτόμο μηχανισμό που υποστηρίζεται και διαχειρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση της υποστήριξης μηνούσμα προς την κοινή δύναμη του G5 του Σαχέλ σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και πάλι το οποίο υπήρξε απαραίτητο γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν για τον σχετικό προϋπολογισμό σε μια επιχείρηση που στην πραγματικότητα δεν είναι επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα ήταν το πρόβλημα, αν θέλετε, τεχνικά της χρηματοδότησης, αλλά βρήκαμε αυτήν τη λύση και θα θέλαμε θερμά να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την για τον ηγετικό ρόλο που ανέλαβε εδώ και την βοήθεια που μας παρήχε. Τώρα η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε με το ταμείο αυτό, όπως και με πολλά ταμεία, είναι ότι έχουμε μια, ένα χρηματοδοτικό κενό. Η Μινούσμα μας έχει πει ότι εντός της αιτίας θα χρειαστεί 44, περί τα 44 εκατομμύρια δολάρια για να παράσχει αυτήν την ε, πολύτιμη βοήθεια στο G5. Μέχρι στιγμής έχουμε είχαμε λάβει μία χορηγία 10 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πέραν της υποστήριξη αυτής της Ένωσης δεν έχει εμφανιστεί κανένας άλλος για να βοηθήσει το οποίο δυσκολεύει την Μινούσμα ιδιαίτερα στην στήριξη που καλείται να παράσχει στα μηχανολογικά στη μηχανική υποστήριξη που παρέχει και που είναι περιοχή ιδιαίτερα κρίσιμη. Ε, η συνολική λοιπόν δέσμη είναι 44 εκατομμύρια των αναγκών, αλλά ε, μας μένει ακόμα, έχουμε πολύ δρόμο για να την καλύψουμε. Και το άλλο που ήθελα να αναφέρω ε, ήταν και η πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την αρχή της πρωτοβουλίας αυτής όπως περιγράφηκε το ψήφισμα 2391 η υποστήριξη προς το G5 και την κοινή δύναμη προχώρησε σε ένα προχώρησε μάλλον εντός πάντοτε ενός πλαισίου πρόνοιας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνεργαστήκαμε στενά με την γραμματεία του G5 και τα κρατημέλη βεβαίως προκειμένου να αναπτύξουμε αυτό το πλαίσιο μέσω στήριξης και ανθρωπίνων πόρων και ο μόνιμος γραμματείας Σιντεκού έχει και αυτός διαγραμματίσει το δικό του ρόλο για να κινητοποιήσει ε, μέλη του G5 ώστε να κινητοποιήσουν τις απαραίτητους μηχανισμούς για ένα πλαίσιο δέουσας επιμέλειας για τους κρατούμενους, για την επιλογή του προσωπικού. Όλο αυτό είναι ένα ευρύτατο πλαίσιο δέουσας επιμέλειας που προχωρεί παραλλήλως προς όλη την υπόλοιπη προσπάθεια και πρέπει να συνεχίσουμε εδώ τη δράση μας σε αυτό το πεδίο χαιρετίζοντα βεβαίω και την ενίσχυση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαριστώντα την. Ευχαριστώ κύριε Κιν. Να δώσω και εγώ κάποιες προφορίες. Η εντολή του G5 εκπνέει όσον ούπο. the format of joint consultation, και η εντολή αυτή δόθηκε μετά από κοινέ διαβουλεύσεις. Υπάρχουν και τα οικονομικά θέματα. Έχουμε τρεις συντονιστές. Ο κ. Γκάλερ πρώτος. German. Θα μιλήσω γερμανικά, οπότε αν χρειάζεστε ακουστικά βάλτε τα σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Ε, και μου έχουν γεννηθεί διάφορα ερωτήματα τώρα. Από τη μια, έχουμε εκεί μια πληθώρα διεθνών δομών στο Μαλή που ασχολούνται κατά κάποιο τρόπο με το να βοηθήσουν τον κρατικό μηχανισμό κάποια στιγμή να αναλάβει τα ενία της χώρας. Όλες αυτές οι δομές λοιπόν που δρούν επί τόπου συντονίζονται Φυσικά με την κυβέρνηση του Μαλή πάντα. Για να μην εργάζονται ο ένας απέναντι στον άλλον. Αν μέτρησα σωστά έχουμε τη Μινούσμα, έχουμε το G5, έχουμε ε, τις εκπαιδευτικές αποστολές. Κάτι ε, άλλο που λεγόταν αφίσμα υπάρχει ακόμα. Έχουμε την επιχείρηση Μπαρκάν από τη Γαλλία. και από διάφορα κράτη-μέλη, ε, απεσταλμένους ειδικού. Προηγουμένως, ακούσαμε για τον κίνδυνο επικαλύψεων και διπλών δομών. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ περισσότερες από διπλές. Έχουν συμφωνήσει. Ποιος είναι ο εχθρός? Ισλαμιστές εντός της χώρας, εκτός της χώρας, από το Μπόκο Χαράμ διεισδύουν και πώς γίνεται η διάκριση των ε, Ισλαμιστών μαχητών από ένοπλους ε, εγκληματίες του κοινού εγκλήματος. Μπορεί να υπάρχουν και ένοπλοι βοσκοί που να φυλάνε εκεί πέρα τις κατσίκες τους και να οπλοφορούν γιατί φοβούνται. Εσείς πώς κάνετε τη διάκριση εκεί, ποιος είναι τι. Και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, Υπάρχει η διευκόλυνση για την ειρήνη αφρικανική που μπορούμε να στείλουμε εκεί χρηματοδότηση. Από εκεί φεύγει πάει στην Άψα που είναι αυτή η αρχιτεκτονική για την ασφάλεια και την ειρήνη. Και αν κατάλαβα καλά, θα σχεδιαστεί μία δύναμη που θα είναι και σε επιφυλακή. Ε, θα φτάσουν εκεί τα χρήματα Κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν ποιος έχει το γενικό πρόσταγμα. Εμένα δεν με νοιάζει. Ας είναι η Μινούσμα. Ε, δεν έχω πρόβλημα. Ή το G5. Αλλά κάποιος να αναλάβει ε, τη διοίκηση και το συντονισμό όλων αυτών που γίνονται. Ε, είναι καλός ο συντονισμός και βέλτιστο το αποτέλεσμα. Πώς το βλέπουν τα μέλη του πάνελ αυτό. Ευχαριστώ η κυρία Λόιζινγκ. Και εγώ γερμανικά θα μιλήσω. Ε, κρατήστε τα ακουστικά σας, παρακαλώ. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Ραζάλη. Το Σεπτέμβριο του 2018, μεταξύ άλλων το Spiegel Online ανέφερε μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ουσιαστικά σφαγές κανονικές μακελιό από το G5 και τη και των χωρών του Σαχέλ. Έκτοτε τι έχει γίνει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ερώτηση προς την κυρία Σνάμπελ. Πώς αξιολογείται τα χρήματα ε, για ε, το στήσιμο του G5 και τη διατήρησή του από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για, για την Αφρική, άρα και από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, το Ταμείο Ανάπτυξη. Ευχαριστώ, η κυρία Βαλέρο. Yes, I I would like to Θα ήθελα να ξεκινήσω με την έκθεση της Γενικής Γραμματείας από πέρυσι, του Ιουνίου του 2018. Κάποιες φράσεις στην έκθεση αυτή, τα μέλη των δυνάμεων ε, ασφαλείας του Μαλή ε, έκαναν 58 παραβιάσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλή υπό, την, ε, υπό το G5 σκότωσαν σε αντίπεινα 5 αμάχους. Ε, η Μινούσμα ε, ερεύνησε σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιτικού Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του Μαλικού στρατού στην περιοχή. Ε, επιπλέον 44 εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και εξαφανίσεις. Όλα αυτά τα ερωτήματα, όλα αυτά τα ζητήματα μας ανάγκασαν να υποβάλουμε ερώτη, ερώτημα στην κυρία Μογκερίνη, στην υπατή εκπρόσωπο, για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να ερευνήσει αυτά τα εγκλήματα πολέμου, αλλά η απάντηση ήταν πολύ συγκεχημένη. Αυτό που θα θέλαμε να καταλάβουμε τώρα είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρακολουθεί τις, τις στρατιωτικές δράσεις και τις πολιτικές αυτές, η BRB, ε, που τις πλαισιώνει υπό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση την νομοθεσία θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση κινδύνου και συνεχής παρακολούθηση. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Πώς ε, παρακολουθούμε τις πολιτικές CBRD ε, και τις ε, στρατιωτικές δράσεις. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα επεισόδια τώρα από κάποιους στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων του Μαλή. Υπάρχει διαφορετικό πρόβλημα εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν για να παρεμποδίσουμε τέτοια επεισόδια και για να μην εμπλέκεται μέσω η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εγκλήματα πολέμου. Δεν θα θέλαμε να μασύρουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επομένως, τι κάνουμε τώρα. Ξέρουμε τι συνέβη. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα για να μην επαναληφθούν τέτοια συμβάντα στο μέλλον. Επίσης, τα εγκλήματα που διενεργήθηκαν ε, τα έχουν εξετάσει όπως πρέπει η, η δικαιοσύνη, τα έχει αντιμετωπίσει όπως πρέπει η δικαιοσύνη του Μαλή ε, και υπάρχει και αποζημίωση των θυμάτων. Τι θα γίνει τώρα. Υπάρχει περίπτωση αναστολής των επιχειρήσεων για τη στήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στείλουμε ένα μήνυμα στον ε, στρατό στι άνθρωπε δυνάμει του Μαλή. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω κάποιε ερωτήσει. Υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία ε, κοινών, ε, μάλλον στρατιωτικής ακαδημίας και αστυνομικής ακαδημίας, κοινών ακαδημιών, για όλη την περιοχή, για τις χώρες όλης τις, όλες τις χώρες περιοχής. σε όλες τις ειρηνευτικές αποστολές υπάρχει και η μη στρατιωτική διάσταση, η πολιτική διάσταση. Και αντίστροφα. Επίσης, τι εξελίξεις έχουμε σήμερα και τι προβλέπετε να γίνει στο μέλλον ε, σε επίπεδο G5. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αστυνομική διάσταση. Τι διαφορές έχει με το στρατιωτικό επίπεδο, με τη στρατιωτική διάσταση. Σε ορισμένες περιοχές βλέπουμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται γρήγορα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια περιφερειακή προσέγγιση, θα πρέπει να κάνουμε και διμερείς προσπάθειες για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας για αυτό το θέμα. I the same order, so Mr. Με την ίδια σειρά, ο κύριος Ραζάνη πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε ένα προς ένα τα ερωτήματα. Και να μην ξεχάσω τίποτα. Για την παρουσία πολλαπλών δυνάμεων και φορέων στην περιοχή. Συμφωνώ ότι η εικόνα δεν μοιάζει πολύ ευανάγνωστη. Συμφωνώ. Ειδικά αν δεν γνωρίζει την κατάσταση στην περιοχή. Είναι μια πρόκληση όχι μόνο για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλους. Δεν θα μιλήσω εξ ονόματος των συναδέλφων του ΟΗΕ, αλλά είναι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε. Θα πρέπει να καταλάβουμε την εικόνα καταρχάς που υπάρχει και να δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Με ποιον μαζί, με ποια εργαλεία. Όπως και να τα ονομάσουμε αυτά. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εικόνα... Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαριστεί λιγάκι, πρέπει να την κατανοήσουμε, να την ε, απλουστεύσουμε λιγάκι. Ο συνάδελφος προσπάθησε να σας πει ότι έχουμε από τη μία την ειρήνη και την ασφάλεια. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε ίσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια καινοτομία για μας αυτή η προσπάθεια σε αυτό το επίπεδο και, και από την άλλη προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την περιοχή και να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της περιοχής. Δυστυχώς, η περιοχή, το Μαλί αλλά και όλη η περιοχή, αντιμετωπίζει ανθρωπιστικές κρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εμπλέκεται πάρα πολύ για να στηρίξει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ε, και χρειάζουν ανθρωπιστική βοήθεια και στήριξη. Ποιοι είναι οι εχθροί τώρα όπως ρωτήσατε. Δύσκολο ερώτημα. Μια από τη στιγμή που άρχισαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις, από τις αρχές του 2000, ε, από την, μέσα αυτό το διάστημα, αυτά 19 χρόνια, άλλαξε άρδινη κατάσταση. Υπάρχει το τοπικό δίκτυο της Αλκάιντα, ε, άλλαξαν όμως μετά τα δεδομένα. Ε, λόγω της ε, φύσης των τοπικών τρομοκρατικών ομάδων που αλλάζουν. Υπάρχει ιδεολογία και ριζοσπαστικοποίηση των ομάδων αυτών, αλλά υπάρχουν και άλλοι ε, φορείς, όπως είπε η κυρία Σνάμπελ, οι οποίοι δρούν τοπικά και με βάση το μοντέλο ζωής. Ε, πέρα από την ιδεολογία και πρέπει να καταλάβουμε και τα τοπικά στοιχεία, ας πούμε, της που χρωματίζουν το πώ δρούν αυτέ αυτές οι ομάδες. Υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα και αυτό συνδέεται με την απουσία της ε, κεντρικής εξουσίας. Δεν μπορεί να εξασφαλίσει φυσικά ούτε δημοκρατική διακυβέρνηση, αλλά είναι το κράτος. Ε, το Μαλί έχει γενικά καλό ρέκορντ σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Τη δεκαετία του 2000 είχε καλή, καλό ρέκορντ ας πούμε. Αλλά υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει αδυναμία διακυβέρνησης. Η κεντρική εξουσία δεν ελέγχει μεγάλο τμήμα της επικράτειας του Μαλή. Εκεί δρούμε λοιπόν για να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση και τις πολιτικές της. Και να υπάρξουν ξανά οι βασικές υπηρεσίες ε, του κρατικού μηχανισμού. Αυτό συνδέεται με την ασφάλεια φυσικά και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε με, τις, ε, ε, με τον εθνικό στρατό, ας πούμε, τις εθνικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση θέλουμε να μπορεί να εξασφαλίζει τις ανάγκες του πληθυσμού όχι μόνο απλώς να στέλνει στρατό, ας πούμε, και αστυνομικούς και εσωτερικές δυνάμεις, δηλαδή. Για να υπάρχει ασφάλεια, όπως σωστά είπατε, εάν υπάρχουν πηγές κατάχρησης, αν υπάρχουν προβλήματα, ε, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια στην περιοχή, στη χώρα. Αυτό θέλουμε να καλύψουμε, αυτό το κενό, ε, εκεί δραστηριοποιούμεθα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ο μηχανισμός ε, για τη χρηματοδότηση της ειρήνης χρηματοδοτεί την, ε, τις προσπάθειες ασφάλειας ε, μαζί με την Αφρικανική Ένωση ε, μέσω της άψα Υπάρχει μια δυσκολία βεβαίως να συνδυάσουμε τα διάφορα εργαλεία που έχουμε για να υποστηρίξουμε την ε, ειρήνη και την ασφάλεια στη χώρα. Σε ό,τι αφορά την Μινουσμά, ε, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εικόνα και η εντολή είναι αρκετά ξεκάθαρη. Γιατί αυτό που κάνει η Μινούσμα δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μόνη μπορεί να το κάνουν είναι αυτή. Δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε το, τη σημασία που έχει αυτή η συγκεχημένη εικόνα. Όλοι μπορούν να βάλουν το λιθαράκι τους. Φυσικά συμφωνώ μαζί σας ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξασφαλίσει κάποιο συντονισμό. Αυτό είναι βασικό της ε, καθήκον ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν συνεργαζόμαστε με τη Μινούσμα, όταν δουλεύουμε τη Μινούσμα, Έχουμε το ψήφισμα 23 91 που παρά την περίπλοκη κατάσταση εξηγεί ποιος κάνει τι. Έχουμε την Αφρικανική Ένωση, υποστηρίζει κάποιες από τις ανάγκες των, της κοινή δύναμης του G5 μέσω της Μινούσμα. Παρότι είναι περίπλοκα τα πράγματα, τελικά ο καθένα ξέρει πολύ καλά τι, θέλει, τι πρέπει να κάνει και τι θέλουμε να πετύχουμε. Πριν περάσω στα άλλα ερωτήματα τώρα, της κυρίας Λόζινγκ, τι γίνεται στο Μαλί. Αυτό που, ό,τι συμβαίνει στο Μαλί δεν παραμένει στα σύνορα της χώρας. Ε, γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να δραστηριοποιήσουμε, να δραστηριοποιηθούμε συγγνώμη, σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει μια, έτσι, ένα φαινόμενο, ας πούμε, χιονοστιβάδα, Ό,τι συμβαίνει στο Μαλί επηρεάζει και τις υπόλοιπε χώρες. Προσπάθησα λοιπόν να απαντήσω στι δικέ σα ερωτήσει, ε, κύριε Γκάλε, κυρία Λέζιν. Ξέραμε τι συνέβη στο Μαλί. Δύο φορές, το οποίο ανέφερε το Σπίγκελ, Η κυρία Μογκερίνη, όπως ξέρετε, αντέδρασε αμέσως και καταδίκασε το περιστατικό και ζήτησε από την κυβέρνηση του Μαλή τι έκανε. ούτω ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα, να γίνει η δικαστική έρευνα και να δοθεί η απαραίτητη συνέχεια. Από ό,τι ξέρουμε, οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχουν ληφθεί πειθαρχικά μέτρα. Τα άτομα από τα τάγματα αυτά, τα οποία έχουμε υπόνοιες ότι έκαναν αυτές τις ε, δράσεις, έχουν, ε, είναι σε, δεν πια, δεν έχουν... είναι σε διαθεσιμότητα δεν ασκούν πια τα καθήκοντά τους. Θα επανέλθω σε αυτό. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και δεν θέλουμε να συρθούμε σε κάτι το οποίο είναι αντιπαραγωγικό. Υπάρχουν καταχρήσεις από τα τάγματα της κοινή δύναμης των G5 και υπάρχουν και καταχρήσεις από τις ε, εθνικές ένοπλες δυνάμεις. Δεν θέλω να πω ότι είναι λιγότερο σημαντικές οι καταχρήσεις του, του G5, αλλά πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Γιατί η άμεση στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς την κοινή δύναμη. Και άρα μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Κυρία Βαλέρο. υπάρχουν αυτά τα επεισόδια στο Μπούλκεση και στο Μόπτι και σε Γκου. Δεν ξέρω αν αυτή η κοινή δύναμη εμπλέκεται. Νομίζω ότι είναι οι εθνικές αναπλές δυνάμεις ε, οι οποίες ε, εμπλέκησαν. Ε, Δεν σημαίνει ότι λιγότερο σοβαρό, λιγότερο προβληματικό αυτό. Αυτό σημαίνει ακόμα περισσότερο ότι πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποια. Και του κράτους δικαίου. Το να φύγουμε από τη χώρα, το να απεμπλακούμε ή το να απειλήσουμε να το κάνουμε, δεν νομίζω ότι θα είναι επικοδομητικό. Θέλουμε η UTM και οι άλλες συνδομές που αναφέρατε, Πρόεδρε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχουν τα, και σέβονται τα επαγγελματικά πρότυπα, ε, ειδικά στο σεβασμό του κράτους δικαίου, τα διοικητικά θέματα, τον τρόπο που μάχονται. Φυσικά, γιατί οι στρατοί πρέπει να αντιμετωπίσουν και την ε, διοικητική πλευρά. Δεν πρέπει να κάνουμε λιγότερα, αλλά περισσότερα έναντι αυτών χωρών και των στρατών τους. Σας είπα τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αναστείλουμε τη UTM. Πρόεδρε. Αυτό συνδέεται και με αυτό που είπε η κυρία Σνάμπελ. Το G5 έχει και εκπαιδευτικές διαδικασίες για την χωροφυλακή, για την αστυνομία και για, και για το στρατό. Κατάρτιση λοιπόν, εκπαίδευση. Και αυτό που κάνουμε και σκοπεύουμε να κάνουμε, στηρίζοντας το G5, αυτά τα μαθήματα θέλουμε να συνεχιστούν λοιπόν. γιατί σε εθνικό επίπεδο υπάρχει έλλειψη δυναμικού. Δεν μπορούν να κινητοποιήσουν στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά δεν μπορούν να κινητοποιήσουν και αστυνομικές δυνάμεις, μη, ε, στρατιωτικέ δηλαδή, πολιτικές δυνάμεις, αστυνόμους, δεν μπορούν να τους βρουν και να τους κινητοποιήσουν. Συμφωνούμε λοιπόν με αυτό που είπατε, ότι το μη στρατιωτικό σκέλος εμπλέκεται πιο πολύ στην ε, κοινή δύναμη Αν εμπλέκεται περισσότερο, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνού δικαίου. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Στάλμαν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Επειδή είμαι ακρηγόρησε σχετικά ο συνάδελφος, θα προσπαθήσω εγώ να είμαι σύντομο. Ε, ε, κατά τα άλλα, απάντησε πολλέ από τι ερωτήσει σα. Να επανέλθω λίγο σύντομα σε ορισμένε ερωτήσεις για τις δομέ συντονισμού και πώς συνδέονται οι διάφορες δράσεις επί τόπου. Για μας ε, όλες αυτές οι αποστολές ε, ε, είναι διαφορετικές. Το G5 έχει δομή συντονισμού ίδια, ξεχωριστή και ήταν συνειδητή επιλογή αυτό. Θα αφήσω να απαντήσει η κυρία Σνάμπελ ε, στην ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και πώς ε, χρηματοδοτεί την Αφρικανική Διευκόλυνση. Ε, πάντως ε, επιλέξαμε συνειδητά σε αντίθεση με άλλες στρατιωτικές αποστολές στην Αφρική να περάσουμε μέσα από το G5 και όχι από την Αφρικανική Ένωση για λόγους καλύτερης λειτουργίας, μονιμότητας ε, και επίσης ε, ιδιοκτησία θα πρέπει να το κάνουν κτήμα του εκεί οι χώρες του G5 γιατί η Αφρικανική Ένωση δεν δραστηριοποιείται πάρα πολύ σε αυτή την περιοχή. Ε, ο συνάδελφος απάντησε διεξοδικά για την εντολή. Η εντολή είναι να αντιμετωπίζει το λαθρεμπόριο και τους εξτρεμιστές που είναι πολύ ευρία έννοια. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την αστυνομία, γιατί όταν ο στρατός συλλαμβάνει κάποιου ε, ε, λαθρεμπόρους ή εξτρεμιστέ, δεν μπορεί να τους δικάζει ο στρατός. Θα πρέπει να περνάνε από τα τακτικά δικαστήρια, με την ε, κανονική οδό, την αστυνομική οδό, ε, μια αστυνομία που δράσει σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και προβλέπεται αυτό και με τη συμπραγματική χρηματοδότηση να προωθήσουμε ε, αυτό ε, ένα σκέλος ε, αστυνομίας πέρα από το στρατιωτικό. Σε ό,τι αφορά τις σφαγή στο Μαλί και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απάντηση που έχουμε να δώσουμε εμείς σε πλευρά ευρωπαϊκή Ένωση ποια είναι. Υποχρεώσαμε το G5 στην κοινή στρατιωτική δύναμη να ενστερνιστεί ε, τα ισχύοντα στα Ηνωμένα Έθνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και θυμίζω, έχουν δεσμευτεί οι στρατοί και οι ένοπλες δυνάμεις των πέντε κρατών. Τι να κάνουν να ελέγχουν ε, τους ε, στρατιώτες, ε, τα βιογραφικά τους, να τους εκπαιδεύουν, να έχουν διαδικασίες για να διαχειρίζονται τις καταγγελίες και να δίνουν συνέχεια και να υπάρχουν έρευνες και δικαστικές και πειθαρχικέ. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο αλλά δεν τον εξαλείφει. Προφανώς και κίνδυνος, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδεθεί με ένα πρόβλημα το όνομά της, ε, δεν είναι ανύπαρκτος, ε, περιορίζεται. Αλλά αυτό το κίνδυνο τον ξέραμε. Ε, θέλαμε από πολιτική σκοπιά να εμπλακούμε, να συνεργαστούμε για το στρατιωτικό σκέλος και το σκέλος ασφαλείας με την ομάδα των G5. Δηλαδή πολιτικά δεν μπορούσαμε να αδιαφορήσουμε, να μην τους πλαισιώσουμε, να μην τους βοηθήσουμε, περιορίζοντας τον κίνδυνο. Και κινδυνεύει και η φήμη φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κύρος της. Αυτή η κοινή δύναμη είναι η πρώτη ε, πολυεθνική αφρικανική δύναμη που έχει ε, εγγραφή σε αυτό το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πρώτη φορά που σημαίνει αυτό, θα μπορούσαν οι συνάδελφοι από το ΟΗΕ να συμπληρώσουν. Και τέλος, για την ε, ε, περιφερική επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, όπως ανέφερε η Πρόεδρος, φυσικά γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στο Μαλί επιδεινώνεται και κυρίως στην Πορκίνα Φάσο με πάρα πολύ ταχύς ρυθμούς. Και έχουμε προβλέψει και επιπλέον χρηματοδότηση διμερή για τις δύο χώρες αυτές και θα πρέπει να αναλύσουμε τη δυνατότητα της κοινή δύναμης αυτής των G5 να ε, δράσει ταχύτατα και στην Πορκίνα Φάσο. Σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να είστε τρίτος ή τέταρτος ομιλητής που καλείται να απαντήσει. Επομένως, ε, κυρία μου ε, και κύριε Κιν, μπορείτε να επιλέξετε από τα θέματα που έθεσαν τα μέλη. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, με μεγάλη χαρά θα το ακούσουμε. Η κυρία Σνάμπελ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τώρα και εγώ γερμανικά. Ήδη υπόθηκαν πολλά. Για τη δική σας ερώτηση, κύριε Γκάλερ, μπορώ να απαντήσω το εξής. Το Σαχέλ είναι ε, πραγματικά πεδίο βολής και ασκήσεων πολλών στρατιωτικών δυνάμεων. Η πρώτη ήταν ε, η ε, Οικονομική Κοινότητα Δυτικής Αφρικής, μετά η Αφρικανική Ένωση και μετά ως ήθιστε τα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί δεν υπάρχουν σε επιφυλακή έτοιμες να επέμβουν πια αφρικανικές δυνάμεις, αλλά είναι θέατρο πολλαπλών ε, συμμετεχόντων, αλλά υπάρχει και πολλαπλή συνεργασία για τη χρηστή διακυβέρνηση κτλ. Και όλα αυτά είναι υπό την αιγίδα της Συμμαχίας του Σαχέλ, ως περιφερειακή αντιμετώπιση που ασχολείται και με θέματα ασφαλείας αλλά και με θέματα ανάπτυξης. Δυστυχώς είναι πολλά ε, τα κομμάτια του παζλ, οι ψηφίδες αυτές ε, που λειτουργούν παράλληλα και δεν υπάρχει συστηματική συνεργασία και συνέργεια. Οι μένα εργάζονται στην αναπτυξιακή βοήθεια και οι δε στην στρατιωτική συνεργασία, αλλά μεταξύ τους δεν υπάρχει ε, συνεπής ε, επεξεργασία ακόμα και των αιτίων της ε, κρίσης. Και αυτό θα είναι και ένα από τα πορίσματα των πέντε γερμανικών Ινστιτούτων που ασχολούνται με θέματα ειρήνης. Επίσης, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο και το κράτος, οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλή, είναι ένας παράγων εκεί από τους εμπλεκόμενους ε, στη σύραξη και ο πολιτισμός δεν ε, εμπιστεύεται καθόλου τη δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων. Αυτά. Τι άλλο. Στην ερώτηση της κυρίας Λέζινγκ έρχομαι τώρα. Για τις μεταφορές πιστώσεων, ε, χρημάτων δηλαδή από το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο και την διευκόλυνση για την Αφρική προς το G5 και για μένα διαφαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς να το πω αξιολογεί πολύ ψηλά την στρατιωτική συνεργασία. Το βλέπουμε και από την UCAP τώρα που έχει αναλάβει και την αντιτρομοκρατική δράση και εκπαίδευση. Και κατά την άποψή μου, να το πω αλλιώ. στο G5 και στο UTM δεν εκπαιδεύουμε απλώς ε, τους G5, αλλά και τον στρατό του Μαλή. Αλλά δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αν θα αποσπάσει δυνάμεις αξιωματικούς και οπλίτες στην κοινή δύναμη του G5 το Μαλή. Εμείς τους εκπαιδεύουμε. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει δεν ξέρουμε, δεν έχουμε λόγο σε αυτό. Ή ποιοι θα παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και με ποια ιδιότητα κάθε φορά αν είναι ε, στρατός του Μαλή ή αποσπασμένοι στο G5 με την υποστήριξη του ΟΗΕ. Λέτε ότι υπάρχει τώρα ένα πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά εκεί παραμένει το ερώτημα της υλοποίησης. Γιατί υπάρχει αστυνομία στη χώρα για να τηρεί την τάξη την οποία καθόλου δεν εμπιστεύεται ο πληθυσμός. Δεν υπάρχουν θεσμοί που να ελέγχουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέρα από τα εθνικά σύνορα. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Thank you. ευχαριστούμε. Ο κύριος Κίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Έχω την πολυτέλεια να είμαι τελευταίος που μιλώ και έχω ήδη ακούσει την σοφία των προηγουμένων. Κάτι επί το οποίο ε, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι, αλλά είναι καλό να το λέμε. κοιτώντας την κατάσταση στο Μαλί και στην ευρύτερη περιφέρεια στο Σαχέλ, πρέπει να εξετάσουμε ποιες είναι οι πολιτικές λύσεις που μπορούμε να υποστηρίξουμε χρησιμοποιώντας την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών, τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της να κάνει. Στο Μαλί προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια διαδικασία συμφιλίωσης και ειρήνευσης θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή μέσω της ε, ούτως αποκαλούμενης Επιτροπής Παρακολούθησης, να δούμε τη διαδικασία της συνταγματικής μεταρρύθμισης, ε, στην ουσία τη διαδικασία της οικοδόμησης κράτους. Αλλά αντιμετωπίζουμε και σοβαρότατες ε, στρατιωτικές προκλήσεις ασύμετρης απειλής, η και ανόκρανη βρίσκονται σε κίνδυνο ε, σε μια περιοχή που ονομάζεται Αγκουλχόκ. Ε, σκοτώθηκαν 10 και των Ηνωμένων Εθνών. 16 ε, τραυματίστηκαν και άλλοι 15 περίπου τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά κατόπιν επίθεσης από τρομοκρατικές ομάδες που επιχειρούσαν να καταλάβουν το στρατόπεδο. Ε, σας δίνω απλώς μια εικόνα, μια γεύση της πραγματικότητας. Δηλαδή, ναι, προσπαθούμε να προωθήσουμε μια πολιτική συμφωνία, αλλά έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν παράλληλα. Χρειάζεται λοιπόν καλή την πίστη όλοι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση και όλοι προς αυτό προσπαθούμε και η, κοινή δύναμη του G5 είναι απλώς ένα από τα κομμάτια του παζλ του ευρύτατου αυτού και περιπλοκού πλαισίου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, επειδή αναφέρθηκαν ήδη, πρώτον, συντονισμός, πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε έναν υπουργικό μηχανισμό συντονισμού, δηλαδή η υπουργοί της περιοχής με τη διεθνή κοινότητα από πίσω τους να τους στηρίζει θα συντόνιζαν την προσπάθεια αυτή και ίσως να φαίνονται συγκεχημένα όλα αυτά, αλλά <clears throat> όχι ακριβώς, γιατί η Μινούσμα προσπαθεί να υλοποιήσει την ε, ειρηνευτική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή εκπαιδεύει τον ε, στρατό, η UCAP ε, τις αστυνομικές δυνάμεις, υπάρχει επιχείρηση Μπαρχάν και το G5 για τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και στα χρηματοδοτικά είναι αρκετά περίπλοκο το τοπίο. Φαίνεται και είναι δηλαδή. Αλλά υπό το ψήφισμα 2391 η μηνούσμα είναι παρούσα στο Μαλί, αλλά προκειμένου να παράσχει οργανωτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις G5 στο Μαλί, χρειάζεται χρηματοδοτική στήριξη για να παράσχει την οργανωτική ή την επιχειρησιακή βοήθεια και τα χρήματα αυτά θα πρέπει να ε, ε, προέλθουν από κάποιον ειδικό πόρο, ειδικό ταμείο κονδύλι. Και βεβαίω η κατάσταση στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αυτή που είναι, είναι δύσκολη. Κανείς δεν προσποιείται ότι πρόκειται για μια ρόδινη κατάσταση εδώ και τα πάμε θαυμάσια. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Υπάρχουν ξεκάθαρα παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι δύσκολο να μιλούμε για πολιτική δέωση επιμέλεια για την ανθρώπινα δικαιώματα. Στην ουσία πρέπει να καλύτερα θα κάναμε να μιλούμε για αποτελεσματική υλοποίηση σεβασμού, πολιτική δηλαδή σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνεργασία με τη γραμματεία του G5 και τη διεθνή κοινότητα, εντός της Μινούσμα έχουμε γραφεία ανθρωπιστικής βοήθειας, που ε, ε, φιλοξενούνται αν θέλετε στην έδρα της Μινούσμα. Έχουμε εξετάσει τα κρούσματα αυτά των ε, εκτελέσεων στις οποίες αναφερθήκατε. Έχουν διεξαχθεί κάποιες έρευνες και τις παρακολουθούμε στενά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και θα συμφωνούσα και εγώ για το EUTM. Δεν νομίζω ότι τίφτα θέμα αναστολής Γιατί το κύριο πεδίο της e UTM είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να περάσουμε απλώς από την κατάρτιση στην επιτήρηση, στην υλοποίηση. Και πρέπει να έχουμε άμεσο σχετισμό μεταξύ των βημάτων αυτών στο έδαφος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ λέει Πρόεδρος. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλα ερωτήματα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για μια πληρέστατη παρουσίαση. Να τους χειροκροτήσουμε παρακαλώ όλοι. Thank you very Ευχαριστώ λοιπόν όλους. Έχω δύο ακόμα ανακοινώσεις. Πρώτον, ότι στην Ολομέλεια του Μαρτίου στο Στρασβούργο 11 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα θα υπάρξει μια δυνατότητα τους πρέσβεις της Πολιτικής Επιτροπής και Επιτροπής Ασφαλείας και Βεβαίως η ΣΕΝΤΕ θα είναι ανοιχτή και σε άλλα μέλη, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Έχουμε πράγματι οργανωτικές δυσκολίες με την συνάντηση της συνεδρίας της 21ης Μαρτίου. Δεν είμαστε βέβαιοι πώς ακριβώς θα πάει το πράγμα. Έχουμε μιλήσει με τις συντονιστές και συνεχίζουμε, περιμένουμε απαντήσεις μάλλον. Θα σας ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα της διαβούλευσης που θα έχουμε και τότε θα σας πω και για τα της επόμενης Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, φορτωμένη σημερινή ημέρα με μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστώ τους διερμηνείς, λέγε ευγενικά η πρόεδρος, ευχαριστούμε και εμείς και τη γραμματεία και όλους εσάς.